Dear colleagues, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ όλους τους προσκεκλημένους μας, τους ομιλητές μας, για τη δημόσια αυτή ακρόαση που έχουμε οργανώσει όσον αφορά τη δέσμη για την τραπεζική νομοθεσία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε. Η ακρόαση αυτή έρχεται πράγματι σε μια πολύ σημαντική στιγμή γιατί ετοιμάζουμε τις εκθέσεις μας για το ίδιο θέμα. Αρχίζει η νομοθετική διαδικασία λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έναν τομέα ο οποίος είναι ζωτική σημασίας για την λειτουργία, ε, για τους κανόνες μας προκειμένου να προχωρήσουμε στην ε, Τραπεζική Ένωση. Αρχίζουμε λοιπόν με μια πολύ καλή βάση πιστεύω και θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση που έχει υποβάλει και στις δύο πλευρές. Η περιγραφή του πακέτου θα ήταν ενδιαφέρουσα. Ίσως θα έπρεπε να ενημερώσω ότι αποφασίσαμε ήδη να προχωρήσουμε σε δύο διατάξεις του πακέτου αυτού, του τραπεζικού, όσον αφορά για παράδειγμα την έκθεση. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα όσον αφορά το fast tracking για τις διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στα άλλα πακέτα, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα και ίσως η συζήτηση αυτή να μας βοηθήσει για να καταλήξουμε. Όπως είπα, τα σχετικά πακέτα έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Η εφαρμογή του TILAC, για παράδειγμα, είναι ζωτική σημασίας, προκειμένου να είναι αξιόπιστη η διαδικασία μας εξυγίανσης η συνολική ικανότητα δηλαδή, απορρόφηση απολειών και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο τέτοιων κανόνων. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτό. Τους επόμενους μήνες, μάλλον την επόμενη χρονιά, θα μπούμε σε έναν περισσότερο σε βάθος προβληματισμό σχετικά με την οδηγία ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών. Γι' αυτό θέλουμε τα δύο στοιχεία να τα αφήσουμε χωριστά. Όσον αφορά τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει, νομίζω ότι υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα αποφυγή κινδύνου και τα μέτρα εκείνα τα οποία δίνουν περισσότερα κίνητρα για καλύτερη διαχείριση στην πραγματική οικονομία. Πάντως, και τα δύο πακέτα και οι κεφαλικές απαιτήσει και η ανάκαυση και εξυγίανση τραπεζών θα βελτιωθούν σίγουρα από το έργο μας και αναμένω η δημόσια αυτή ακρόαση να προσφέρει περισσότερα στοιχεία προβληματισμού προκειμένου να προσφέρουμε και εμείς έργο υψηλής ποιότητας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους εισηγητές μας πρώτα απ' όλα για πέντε λεπτά ο καθένας παρακαλώ και πρώτα για το πακέτο όσον αφορά την ανάκαμψη εξυγένσης ε, και εξυγένσης τραπεζών, ο κύριος Χόκμαρ. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή και θέλω και εγώ να καλωσορίσω εδώ τους σημερινούς μας προσκεκλημένους. Από την δικιά μου την πλευρά θα αρχίσω λέγοντας ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια περάσαμε από μια πολύ σημαντική διαδικασία εκπόνησης νομοθετικού έργου στον τομέα αυτό. Οι κεφαλικές απαιτήσει, η οδηγία και ο κανονισμός είναι το ένα στοιχείο, η οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών είναι ένα άλλο και έχουμε και άλλα ζητήματα πάνω στα οποία έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι ρυθμίσεις για την διαθέτηση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Τώρα αναλαμβάνουμε ένα παραπάνω βήμα προς τα μπρος, γιατί έχουμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε το τι πετύχαμε μέχρι τώρα και πού παραμένουν προβλήματα. Είναι λοιπόν θετικό να ακούσουμε τους διαφορούς ομιλητές για να δούμε πώς προχώρησε η εφαρμογή των κανόνων αυτών, ποιες είναι οι εμπειρίες μας από τα διάφορα αυτά νομοθετικά πακέτα που έχουμε γκρίνει μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, όσον αφορά την οδηγία ανάκαμψη και εξυγένση τραπεζών, η BRRD, δοκιμάζεται σε μερικέ περιπτώσει. Καλό θα ήταν λοιπόν να ακούσουμε εμπειρίε πάνω σε αυτό. Επίση, να ακούσουμε πώ η νομοθεσία αυτή έχει εφαρμοστεί στι διάφορε χώρε μέλη. Ίσως τα προβλήματα να έχουν να κάνουν και με διαφορετικές μορφές εφαρμογής και υλοποίηση των όσων προβλέπονται σε αυτή την οδηγία. Πάντα λοιπόν για την οδηγία ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών ένα σημαντικό στοιχείο είναι να επιμείνουμε στην πειθαρχία στις αγορές. Ακριβώς αυτή την πειθαρχία θέλει να προσφέρει η οδηγία BRRD. Οποιοςδήποτε επενδύει σε μία τράπεζα πρέπει να γνωρίζει ότι τα χρήματα, το παθητικό τελικά μπορεί να καλυφθεί ιδίς μέσης, αν χρειαστεί. Πρέπει δηλαδή να δούμε ποιο είναι, ποιες είναι οι δυνατότητες επίσης που προσφέρει ο εποπτικός μηχανισμός στην Ευρώπη και να γνωρίζει κάθε επενδυτή τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Γιατί ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε διαπιστώσει όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη της οδηγίας ανάκαψης και εξυγίανσης τραπεζών είναι ότι οι αποταμιευτές θεωρούν ότι το κεφάλαιό τους δεν διασφαλίστηκε όπως έπρεπε, ενώ στην πραγματικότητα αυτό έγινε. Και αυτό είναι που πρέπει να βγει από αυτή τη διαδικασία. Να διευκρινίσουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Επειδή μέρος του χρέους, μέρος του κεφαλαίου σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο που να επιδέχεται περισσότερο διάσωση δις μέσης από ότι ένα άλλο κομμάτι του ίδιου κεφαλαίου, του ίδιου χρέους. Και τι γίνεται και με το κεφάλαιο. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε ένα από τα πράγματα που με μεγάλη αποφασιστικότητα θελήσαμε να διασφαλίσουμε όταν σχεδιάσαμε την οδηγία ανάκαμψης και εξυγένσης τραπεζών. Θέλω λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από αυτόν. Η εισαγωγή τώρα του TILAC στο σύστημα αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζουμε ότι το χρέος μπορεί να ε, διασωθεί οι δύο μέσης γρήγορα και να μην δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν άλλα τμήματα ε, του χρέους μιας τράπεζας που δεν διασώζεται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Επίση, ζωτική σημασία είναι να δούμε και τα διάφορα αυτά θέματα σαν στοιχεία ενός συνόλου. η οδηγία δηλαδή και ο κανονισμός για τις κεφαλικές απαιτήσει μαζί με την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίαση τραπεζών. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και έχουμε συζητήσει το πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία εγώ με τον κύριο Στήμαν, ο οποίος είναι συγκητής για το άλλο κομμάτι του πακέτου και είμαστε πραγματικά αποφασισμένοι να πετύχουμε. Αυτό που επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι προχωρώντας με κοιτάτε σαν να έχω ξεπεράσει τον χρόνο μου. Εντάξει, 10 δευτερόλεπτα δώστε μου. Τα έχω εξάλλου. Ναι, πειθαρχία, ναι, ναι, είπα πειθαρχία αγορά, σύμφωνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει ούτε ο πρόεδρο να υπονομεύει την πειθαρχία τη αγορά. Λέει ο κύριο Χόκμαρ. Και συνεχίζει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να προσφέρει σταθερότητα, συγχρόνω όμω με δυναμισμό στα χρηματοπιστωτικά στι αγορέ μα. Οπότε, με 25 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, τα οποία ταξόδεψα όταν με κοιτάξατε με αυτό το βλέμμα πριν, τελειώνω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ισηγητά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες ε, στην ε, σημερινή μας ακρόαση. Παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας και να αφαιρέσετε το χρόνο αυτόν από το χρόνο ομιλίας μου. Να μηδενίσετε δηλαδή το ρολόι πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, διότι οι δέσμοι νομοθετικών μέτρων για τις τράπεζες είναι αδιαμφισβήτητα κάτι πολύ σημαντικό. Ε, βασίζεται σε αποφάσεις ε, της Βασιλείας και έχουμε έτσι νομοθετικές και τεχνικές καινοτομίες ε, τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Βρισκόμαστε σε μια φάση προσανατολισμού. Με μεταβατικές διατάξεις για το ISF 9 μπορούμε με ξεχωριστή μεταχείριση του ISF9 μπορούμε να μικρύνουμε την μεταβατική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που βρίσκεστε εδώ σήμερα και ως εισηγητής έχω εντοπίσει κάποια θέματα τα οποία θεωρώ ότι ε, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό και γι' αυτό θα θέσω συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα διότι κατά τη διάρκεια της ακρόασης δεν θα έχω τη δυνατότητα να θέσω ερωτήσεις. Καταρχάς, είσαι συνθήκες ανταγωνισμού και αναλογικότητα. Πρέπει να έχουμε ομοιόμορφους κανόνες, αλλά αυτό είναι δύσκολο στην ε, ποικιλόμορφη ευρωπαϊκή αγορά. Ε, κάποια ιδρύματα θα πληγούν δυσανάλογα από τις νέες ρυθμίσεις. Ε, άλλοι οργανισμοί δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς και θα οδηγηθούν σε συγχωνεύσεις. Έχω εδώ ένα άρθρο από την Frankfurter, Frankfurter Allgemeine Zeitung ε, όπου βλέπουμε ότι κάποια, κάποιοι οργανισμοί που πρέπει να κλείσουν είναι ε, θύματα αυτού του νομοθετικού τσουνάμι, γράφει η εφημερίδα. Πώς ε, βλέπετε εσείς λοιπόν τις προτάσεις της Κομισιόν υπό το φως της αναλογικότητας. Ε, πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και επίσης που πιστεύετε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ελαφρύνσεις και παρεκκλήσεις πέρα από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Επίσης, Όσον αφορά την, ε, τον έλεγχο των κινδύνων, ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ε, αυξάνονται οι απαιτήσει με το μέγεθος και Επίσης έχουμε τον κύριο Τράιχελ και άλλους δύο Αυστριακούς ομιλητές εσείς εκπροσωπείτε μικρές τράπεζες. Τι δυνατότητες πιστεύετε ότι υπάρχουν για ελαφρύνσεις για τα μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα με ενδιαφέρε να γνωρίζω ε, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ε, που δημιουργούνται από την οδηγία και τον κανονισμό για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις, CRR και CRD. Επίσης, ε, από τον εκπρόσωπο της Societe Generale θα ήθελα να ακούσω γενικά υπάρχουν κάποια ε, εσωτερικά σχέδια ε, και οι μικρομεσαίες τράπεζες χρησιμοποιούν μία σειρά πρότυπων κανόνων. Εσείς, λοιπόν, τι περιορισμούς πιστεύετε ότι θα επιβάλλει το πρόβλημα αυτό των κινδύνων και επίσης ποια θέματα είναι ασύμβατα με συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Πώς πιστεύετε, ποια, ποιοι κανόνες πιστεύετε ότι θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους μεγάλους οργανισμούς. Η αναλογικότητα λοιπόν και οι συνθήκες ίσου ανταγωνισμού είναι θέματα πολύ σημαντικά για μένα και από τους εκπροσώπους των τραπεζών ακούμε όλο και πιο συχνά τα ίδια στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την EBA και άλλους. έχω ακούσει την άποψη. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κεντρική αρχή όπου να διαβιβάζονται όλα τα σχετικά δεδομένα και ο χρήστης να μπορεί να αναζητήσει εκεί τα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν. Για τέτοια ενοποίηση των δεδομένων ε, θα αποτρέψει την ε, επικάλυψη των εργασιών ε, και θα διασκεδάσει και τις ε, αμφιβολίες. Εσείς πώς βλέπετε την ιδέα αυτή. 5 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, όπως και ο κύριος Χέκμαρ. Ε, και, και μάλιστα χωρίς να με αγροκοιτάξει και ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις. Θα ακούσουμε τους ομιλητές μας. Αντρέα Ανρία Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζική Αρχής. Καλώς ήρθε, Ανδρέα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η υπηρεσία μου καλωσορίζει την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστούν διεθνεί προδιαγραφέ στο εθνιστικό πλαίσιο. Συμβάλαμε στι προτάσει μέσω σειρά εκθασών για το ποσοστό μόχλευση, ποσοστό χρηματοδότηση, ελάχιστε απαιτήσει ε, για τι διάφορε ε, ευθύνε Διεξοδικά αναλύσαμε τα αποτελέσματα τη εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών στι ευρωπαϊκέ αγορέ. Εξολογήσαμε τι συνέπειε που έχει για διάφορα μεγεθά πεζών, για υπηρεσιακά μοντέλα και δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όσον αφορά εν γέννη την ευρωπαϊκή οικονομία. Η σύστασή μα ήταν να ευθυγραμμιστούμε με τι διεθνεί προδιαγραφέ με μικροπροσαρμογέ και χαιρόμαστε που οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη έχουν αποδεχθεί τα συμπεράσματά μα. Υπάρχουν μόνο μερικοί τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάπω ξεφεύγει από τι διεθνεί προδιαγραφέ και από τι θέσει τι δικέ μα. Ε, χαλαρώνονται οι απαιτήσει για κάποιε συναλλαγέ σε ε, συγκεκριμένου οργανισμού. Αυτέ οι προτάσει διατηρούνται στο τελικό κείμενο. Αν μείνουν, θα πρέπει να δοθούν εντολέ στην υπηρεσία μα να παρακολουθεί τα διάφορα προβλήματα και να υπάρχει συντηρητική εφαρμογή όλων των εξαιρέσεων σε όλη την ενιαία αγορά. Ε, ένας από τους στόχους του πακέτου είναι οι κανόνες ε, του CRD και του CRR να γίνουν πιο αναλογικοί. Όπως έλεγε ο Σίμων, ε, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τα ιδρύματα με μεγάλο άχθος. Ζητά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ρυθμιστικό πλαίσιο για τι χρηματοπιστικέ υπηρεσίε. Χρειάζεται να δούμε ποιο είναι το βάρο τη συμμόρφωση για τι μικρέ υπηρεσίε με ένα ενιαίο επιχειρηματικό μοντέλο με παραδοσιακέ συναλλαγέ. Το κόστο τη υποβολή αναφορών, και αν θέλουμε να έχουμε περισσότερες απαιτήσει στο κοινό πλαίσιο αναφορών είναι κάτι που μας ανησυχεί. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι η αναλογικότητα στις ρυθμίσεις περί τραπεζών ε, είναι κάτι που υπερέχει των λιγότερων απαιτήσεων για τις τράπεζες. Οι ρυθμιστικές απαιτήσει δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με τους κινδύνους. Όχι αυτό θα πρέπει να υπάρχει αναλογική εφαρμογή των κοινών κανόνων. Χρειάζεται εξορρόπηση ομοιομορφών κανόνων με διαφοροποίηση συμμορφώσεων. Έτσι αντικατοπτρίζεται ο περίπλοκο χαρακτήρα και κίνδυνη του πεζικού τομέα. Θα μέσω απλουστευμένη εφαρμογή των κανόνων μπορούμε να έχουμε καλύτερη προσέγγιση και να μειώσουμε το άχθο χωρί να υπολοιπόμεθα των στόχων που έχουμε για συνετή διαχείριση. Άλλο θέμα είναι το θέμα του πυλώνα 2 ε, καλωσορίζονται οι συστάσεις. Καταλάβαν πολύ γρήγορα ότι η παρούσα εφαρμογή των απαιτήσεων του, κανόν, του πυλώνα 2 είναι ποικιλόμορφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντικατοπίζουν μεγάλο βαθμό την άποψή μα που εκφράζουμε στην γνωμοδότησή μα, ε, λόγω τη εμπειρία που είχαμε από τα πρώτα χρόνια εφαρμογή του CRD. Λοιπόν, η πρόταση διευκρινίζει τη φύση και τη μορφή του πυλώνα και των απαιτήσεων αυτού, που είναι δεσμευτικέ απαιτήσει, πρέπει να επιβάλλονται με νομοθετικά δεσμευτικό τρόπο. Διευκρινίζεται η λειτουργία των κανόνων για ε, μέγιστο ποσό αναδιάθεση, ανακατανομή και κάποιε κατευθείαν γραμμέ για τι κεφαλαϊκέ ανάγκε, ούτω ώστε να έχουμε σωστέ προσδοκίε όσον αφορά του ελέγχου, όσον αφορά το κεφάλαιο για τι δοκιμέ αντοχή και ενδεχόμενε απώλειε και συνθήκε δοκιμών αντοχή ε, η χρήση των αποτελεσμάτων ε, δοκιμών αντοχή από τι αρμόδιε αρχέ ε, δεν είναι ομοιόμορφο εφαρμόζοντα ε, τι διάφορε διαδικασίε αξιολόγηση και εποπτεία. Κάποιε αρχέ χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχή για να δημιουργήσουν κατευθυντήρε γραμμέ για τι κεφαλουχικέ απαιτήσει. Άλλε χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών ω δεσμευτικέ απαιτήσει του πυλώνα 2 ή σαν εποπτικά όρια. Τελικά η πρόταση διευκρινίζει τις, τις όσον αφορά τη συνετή διαχείριση για την επιτεύξη μεγαλύτερη σύγκληση όσον αφορά την εποπτική πρακτική που ακολουθείται. Καλωσορίζουμε και τα ψηφίσματα, τις στοιχείες ψηφισμάτων της Πρωτεύουσα Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντικατοπτρίζουν εν γέννη την έκθεση που δημοσιεύσαμε το Δεκέμβριο του 2016, ευθυγραμμίζονται με το, ε, απαιτήσει Τίλα και FSB για τον πυλώνα να πω και κάτι άλλο, ανταποκρινόμενο σε αυτά που είπε ο κ. Χόκμαρ. Είναι σημαντικό ε, να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση PRD για τη διαχείριση των κρίσεων. Ε, απομακρυνόμαστε από το bailout και εσωτερικεύουμε τις απόψεις μέσω ε, διασώσεως από ιδιωτικούς επενδυτές με ίδια μέσα. Αυτή η προσέγγιση μεταξύ άλλων βρίσκεται στη διάταξη ότι αν ένα θεσμικό όργανο χρειάζεται κρατική ενίσχυση, αυτό το θεσμικό όργανο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μπορεί να χρεοκοπήσει, είναι πιθανό να χρεοκοπήσει, αν ε, προκαταρτική κεφαλοποίηση με δημόσια χρήματα είναι εξαιρετικό μέτρο όταν όμως πληρούνται αυστηρές συνθήκες και προϋποθέσεις. Πρόσφατα υπέβαλα μια πρόταση χρησιμοποιήσουμε την αρχή της ε, προληπτικής κεφαλοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να, για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τροπιστικός τομέας. Ε, που δημιουργεί προβλήματα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πρώτα, να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή εταιρεία που διαχειρίζει τα στοιχεία ενεργητικού, χρησιμοποιώντα επίση και εθνικά συστήματα διαχείριση στοιχείων ενεργητικού για να αποτυχούν χρεοκοπήσει και να επιληθούν τα διάφορα προβλήματα. Ε, λοιπόν, πρέπει να σεβόμαστε τις προϋποθέσεις του BRD και έτσι θα πετύχουμε συνοχή στην ενιαία αγορά για σωστή εφαρμογή των κανόνων. Και πρέπει να δράσουμε δυνάμει αυτού του πλαισίου για να είμαστε αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι όσον αφορά την προσέγγιση του συστήματος BRD. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ένδρια. Ντανιέλ Νουή τώρα, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενίου Εποπτικού Μηχανισμού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή τροποποίηση του πακέτου έρχεται την κατάλληλη στιγμή και είναι κάτι αναγκαίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε ισχυρές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις διεθνώς και να λάβουμε υπόψη μας και την πρόεδρο που έχει συμβεί στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ευχαριστούμε που έρχονται τώρα οι προτάσεις αυτές που θα ενισχύσουν την αντοχή των ευρωπαϊκών ε, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ευχαριστούμε για τις αλλαγές που προτείνονται επίσης όσον αφορά την εφαρμογή του TILAC για παράδειγμα, την αναθεώρηση επίσης του πλαισίου MREL που είναι πράγματα που πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Έπειτα, ευχαριστούμε και για την εισαγωγή εναρμονισμένων κατηγοριών μη προτιμησιακών ε, παλιών ε, χρεών που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις νέες απαιτήσεις. Πιστεύουμε επίσης ότι πέρα από την τρέχουσα πρόταση, η προτιμησιακή ρύθμιση για τις καταθέσεις πρέπει όντω να ε, εισαχθεί και να συμπεριληφθεί και το στοιχείο του Μπέιλιν. Ακτιμούμε επίσης τις διατάξεις εκείνες που θα διευκολύνουν την προληπτική εποπτική διαχείριση, ιδιαίτερα για τρίτες ε, χώρες που έχουν ε, τράπεζες στην Ευρώπη. Χρειάζονται κάποιες επίσης τροποποίησεις για να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά το αρμπιτάζ. Σημαίνει ότι η ε, μητρική εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει τις θηγατρικές με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται ε, συγκρούσεις. Τέλος, στηρίζουμε την πρόταση για εξαιρέσεις όσον αφορά το κεφάλαιο, ιδιαίτερα για περιπτώσεις διασυνοριακές. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει πιο αποτελεσματική διαχείριση ε, διασυνοριακά του κεφαλαίου και θα βοηθήσει περισσότερο στην ε, ολοκλήρωση και στην εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς να υπάρξουν στρεβλώσεις όσον αφορά τη σταθερότητα. Βέβαια παραμένουν 7 ε, σημεία όπου μπορεί να υπάρξει παρεντέρω βελτίωση. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι επόπτες διαθέτουν τα μέσα που χρειάζονται όσον αφορά τις αναφορές που κάνουν στη συνέχεια και να συμπεριλάβουν στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο. Όλες οι καταστάσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν από τον πυλώνα 1. Γι' αυτό οι επόπτες χρειάζονται ένα βαθμό διακριτικής ευχέρειας προκειμένου να παρουσιάσουν τα πορίσματά τους. Η πρόταση λοιπόν για το Pillar 2 προσπαθεί να πετύχει μεγαλύτερη σύγκληση σε πολύ βασικά στοιχεία. Η αξιολόγηση του κινδύνου στον πυλώνα 2 θα μας ε, επιτρέψει να έχουμε το κατάλληλο χρηματοοικονομικό αναφορικό πλαίσιο όπου οι επόπτες δεν θα διαφοροποιούνται όσον αφορά τους κινδύνους και όπως αυτοί εξελίσσονται. Είναι επίσης αναγκαία να διασφαλίσουμε ότι οι επόπτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την προσθήκη κεφαλαίου λαμβάνοντα υπόψη τη δυνατότητα απορρόφησης. Έχουμε ήδη εμπειρίες από τέτοια ζητήματα στον πυλώνα 1. Η πρόταση δεν προσφέρει επίσης εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζονται παραπάνω στοιχεία για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα όσον αφορά το κεφάλαιο και να μπορέσουμε προληπτικά να τα αντιμετωπίσουμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα στους κανόνες. Στην περίπτωση μη εξυπηρετούμενων δανείων, για παράδειγμα, που δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εξέλιξη νέων NPS. Τώρα, όσον αφορά την απόκληση από τα διεθνή πρότυπα, εδώ χρειαζόμαστε παρετέρω ανάλυση. Μέχρι τώρα η απόκληση αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη να προσαρμόσουμε τους κανόνες στην ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα, χωρίς όμως να απλήξουμε την αποτελεσματικότητα των κανόνων. Υπάρχουν πολλές διατάξεις που δεν πετυχαίνουν ακριβώς αυτό το στόχο όσον αφορά τις αποκλήσεις από τα διεθνή πρότυπα. Ακόμα και για την επιτυχία της μεγαλύτερης αναλογικότητας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως θέλουμε. Όμως προτιμάμε όχι τη συχνότητα, αλλά την πυκνότητα granularity. Χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία για αναρμόνιση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Μπορούν να γίνουν περισσότερα στον τομέα της εναρμόνισης αυτής. Είναι επίσης σημαντικό ο νομοθέτης να φροντίσει για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Τέλος, είμαστε υπέρ της διευκρίνησης έγκαιρων μέτρων που θα βοηθήσουν τον ε, κάθε επόπτη προκειμένου να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό στο έργο του. Yes. Ε, το χρόνο μου, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δομινίκ Λαμποριέ. Από το Συμβούλιο του ε, Συμβουλίου του Ενιαίου Μηχανισμού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που με κάλεσαν ε, σήμερα εδώ να ε, συμμετάσχω στην συζήτηση για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Μα ακούτε καλά τώρα? Ωραία. 15 δευτερόλεπτα σπατάλησα. Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα να περάσω κατευθείαν στο περιεχόμενο της παρέμβασής μου που θα επικεντρωθεί ε, σε θέματα εξυγίανσης και όχι εποπτείας. Επικροτούμε την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, του MRL και του TILAC και θα θέλαμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολλή δουλειά που έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρινίζει πώς θα εφαρμοστεί το διεθνές πρότυπο ΤΙΛΑ και τη συνολική ικανότητα απόρρευσης απολειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ε, προτινόμενη εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε στο MRL ένα κομμάτι στον πυλώνα 1 και επιπλέον απέτηση του πυλώνα 2. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τις ε, μεγάλες διαφορές ε, ανάμεσα στις ε, μικρές και τις μεγάλες συστημικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα την σημασία του να υπάρχουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού και για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Είναι Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Και γι' αυτό μας αρέσει η σύσταση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ε, να ε, επεκταθεί και σε άλλα συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, η απέτηση του πυλώνα 2 και θέλουμε αυτό να γίνει και για τον πυλώνα 1. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι χρήσιμο ε, κατά τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω στο θέμα αυτό. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρηθεί τουλάχιστον η υπάρχουσα ευελιξία, ώστε η ποιότητα, ο τόπος και τρόπος ε, εφαρμογής ε, των ε, ελάχιστων απαιτήσεων ε, να αντιστοιχεί στις ανάγκες των τραπεζών. Όσον αφορά τα GSIP στις ε, συστημικές τράπεζες, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφώνεται με διεθνείς απαιτήσεις τουλάχιστον την 19 και 22. Όσον αφορά το MRL, η απαραίτητη ευαλιξία για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να δώσει την απαραίτητη ισορροπία δεδομένων των κινδύνων μιας παρατεταμένης μεταβατικής περίοδου. Όσον αφορά την ιεράρχηση των επιστώσεων, όπως ε, ε, επικροτούμε το ότι δίνεται προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Χρειάζεται βεβαιότητα όσον αφορά τα θέματα δανείων. Είναι σημαντικό η πρόταση αυτή να είναι αρκετά στιβαρή και να μην υπάρχουν αμφισημίες. Και όσον αφορά το μορατόριο και τη σχετική πρόταση, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το πεδίο εφαρμογής, διότι υπερβολικά ε, στενό ε, πεδίο εφαρμογής ε, θα καταστήσει το μέσο αυτό άχρηστο, ενώ το υπερβολικό πεδίο εφαρμογής, το υπερβολικά ευρύ πεδίο εφαρμογής θα οδηγήσει σε άλλα προβλήματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μετά από ένα εποπτικό μορατόριουμ είναι δύσκολο για μια επιχείρηση να επιστρέψει στην αγορά, διότι είναι δύσκολο να μην περάσει μετά σε διαδικασία εξυγίανσης. Θα θέλαμε επίσης να εισάγουμε μια γενική ρήτρα για ε, ε, τις εξουσίες αναστολής. Επίσης, Στηρίζουμε την πρόταση για την ενδιάμεση γονική επιχείρηση και έχουμε ε, σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που στηρίζει την πρόταση αυτή. Γενικά, εάν εφαρμοστεί σωστά η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι τράπεζες ε, θα γίνουν πιο ε, ανθεκτικές και αυτό θα ωφελήσει την οικονομία στο σύνολό της. Είναι σημαντικό να μην αποδυναμώσουμε το πλαίσιο που έχουμε σήμερα. Αντιθέτω, θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία που μα δίνει η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε περαιτέρω το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ακούσουμε εκπροσώπους εθνικών εποπτικών αρχών. Έρικ Φιντίν, Γενικός Διευθυντής Φινάς Εξυπηρεσιών που είναι η Σουηδική Εποπτική Αρχή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Σα ευχαριστώ που μας προσκάλεστε μαζί συναδέλφου εδώ στι Βρυξέλλες για να σταθούμε επί της νέα νομοθεσίας περί τραπεζών. Ξεκινώντας να εκφράσω την εκτίμησή μου για το επιτελεστέν έργων. Έργο που ετέλεσε το Κοινοβούλιο για την επιδιώθωση του συστήματο τραπεζικού. Εννέα χρόνια μετά από την κρίση, οι ευρωπαϊκέ τράπεζε έχουν καλύτερη κεφαλοποίηση από όταν ε, μα έπληξε η κρίση. Υπάρχει καλύτερη κυβέρνηση και έχουν μεγάλα βήματα προόδου για μεγαλύτερη εντοχή των τραπεζών. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τέλο του ταξιδιού μα για να διορθώσουμε το τραπεζικό σύστημα. Ζητώ συγγνώμη. Σημαντικέ ρυθμιστικέ ε, ρυθμίσει απαιτούνται και ένα από αυτά είναι το πακέτο αυτό τραπεζικό πλευρά Σουηδία. Καλωσορίζουμε την νομοθεσία αυτή, το πακέτο αυτό, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα όρια που τίθενται όσον αφορά την εποπτική ευελιξία και κυρίω τη δυνατότητα η υποπτική αρχή είναι να αντιμετωπίσει συστημικού κινδύνους και επαναλαμβάνω συστημικούς κινδύνους διότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για την σουηδική περίπτωση. Αυτό, πρέπει να προτείνει κάτι τέτοιο το νομοθετικό πακέτο. Τώρα θα στραφώ προς την πρώτη μου διαφάνεια που βασικά αναφέρεται στα σημεία που θα πρέπει να εξετάσουμε. Να δούμε πώς χρειάζεται ευελιξία, συνύπαρξη ευελιξίας και εναρμόνιση. Η εναρμόνιση καθορίζει ελάχιστε προδιαγραφές δίδει μια προβλεψιμότητα και υπάρχει και μια συνεπής αντιμετώπιση του κινδύνου. Άρα είναι ένας τρόπος ε, αποφυγής ρυθμιστικής διαιτησίας και να αποφύγουμε μια προς τα, τα κάτω προσέγγιση. Και η ευελιξία είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για να εξασφαλίζεται ολιστική αντιμετώπιση και εντοπισμό του κινδύνου, να υπάρχει σωστή στάθμιση των εργαλείων και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι για συγκεκριμένη περιοχή ή για χώρα. Ευελιξία λοιπόν. Και αυτή δημιουργεί κινδύνους. Μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί, βλέπετε, την ευελιξία για εθνικά κέρδη. Το κόστος αυτού όμως είναι πολύ υψηλό και δημοσίας φύσεως και αυτός ο κίνδυνος καμιά φορά έχει τονιστεί υπερβολικά στη συζήτηση. Σας δείχνω κάποια γραφήματα. Βλέπετε ότι η Σουηδία ξεχωρίζει, αλλά και οι άλλες χώρες ξεχωρίζουν και γι' αυτό και το ευρωπαϊκό σύστημα τραπεζικό είναι ποικιλόμορφο. Υπάρχει διαφορετική εφαρμογή του πυλώνα 2. Ίσως δεν είναι κακό, αλλά ίσως αντικατοπτρίζει και την πραγματικότητα. Η Σουηδία έχει το μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα, η συγκρίση με το ΑΕΠ τη μαζί με την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σύγκριση με τη γειτονική μα χώρα στη Φιλανδία έχουμε τριπλάσιο μέγεθος όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα. Διπλάσιο από ότι το Βέλγιο. Άρα, η κίνδυνη στο σουηδικό σύστημα, η συστημική κίνδυνη εξορισμού είναι μεγαλύτερη. Επίσης, εξαρτώμεθα κατά πολύ από τη χρηματοδότηση του τομέα χονδρικής Άρα χρειαζόμαστε εύρυθμη αγορά, λειτουργία αγοράς ομολόγων. Και εκεί βέβαια υπάρχουν συστημική σημασία κίνδυνοι. Και κάτι άλλο που συζητήθηκε εκτεταμένα. Ε, λοιπόν, ε, είδαμε μεγάλη ανάπτυξη στην ιδιωτική δανειοδότηση μαζί με αύξηση των τιμών για τη στέγαση. Και βλέπουμε ότι η Σουηδία που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο έχει αυτή την εικόνα ίσως σε κάποια φάση αυτή την εικόνα θα παρουσιάζει άλλη χώρα. Άρα όμως με αυτό το γράφημα βλέπουμε ότι χρειάζεται ευελιξία. Τι σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να εξετάζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι ε, και υπάρχουν διατερότητες νομικές και περιοχών και χρειάζεται ευελιξία την αντιμετώπιση των κινδύνων. Έτσι θα χειριζόμαστε καλύτερα την κρίση για κάθε κράτος μέλος. Αλλά ο κίνδυνο διάδοση προβλημάτων είναι κάτι που αφορά τα κράτη-μέλη. Τέτοια μέτρα για αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων μπορεί να συζητηθούν σήμερα μέσω συστημικών με, μεταξύ συμπληρώσεων κεφαλουχικών και μέσω μέτρων του πυλώνα 2 που εφαρμόζουμε εκτεταμένα και η προτινόμενη αυτή η νομοθεσία μειώνει αυτή τη δυνατότητα και νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλό ε, για την ε, αντιμετώπιση χρηματοστικών κινδύνων στη Σουηδία και συνεπώς δεν είναι καλό και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η ευελιξία και η εναρμόνιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Θα διερωτάστε τι είναι αυτή η εικόνα που σας δείχνω τώρα. Υπάρχει παραλληλισμός με διαφορετικές συνθήκες καιρικέ στην Ευρώπη, αν παραλληλήσουμε με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τραπεζών. Διαφορά καιρού, διαφορά συστημάτων τραπεζικών. Στη Σουηδία, υποχρεωνόμεθα διανομοθεσίας, να έχουμε λάστιχα από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου να έχουμε χειμερινά λάστιχα. Δεν υπάρχει μέγιστη εναρμόνιση όσον αφορά τα ελαστικά και αυτό έχει, ζώσει, έχει σώσει ζωές. Το ίδιο ισχύει, υπάρχει παραλληλισμός και με την τραπεζική νομοθεσία, αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι εδώ την Ελίζα Φερέιρα μας έχεις λείψει, Ελίζα. Ξέρω όμως ότι δουλεύει σκληρά ως μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών της ε, Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Και νομίζω ότι θα με πιστέψετε όλοι σας όταν με ακούτε να λέω πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου όλων αυτών των χρόνων στο Διευθυντικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Πορτογαλίας. Συμμετέχω στο Εποπτικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει Ντανιέλ επίσης. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι η Τραπεζική Ένωση οικοδομήθηκε πάρα πολύ σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αδιαφεσβήτητα όμως είναι επιτυχία. Θέλω να κερδίσουμε χρόνο εδώ και Ντανιέλ και Αντρέα και Ντομινίκ και άλλοι και τα μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω και της Επιτροπής αυτής, να σας ευχαριστήσω όλους για την επιτυχία αυτή στην Τραπεζική Ένωση. Όμως η τρέχουσα αναθεώρηση των ε, νομικών θεσμών είναι μια ευκαιρία να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Υποφελούμεθα από την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα και είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιοι κρίκοι στην αλυσίδα που εξακολουθούν να λείπουν και κάποια σταθεροποιητικά στοιχεία ε, τα οποία χρειάζονται και για τα οποία πολλές φορές μιλήσαμε εδώ είπατε πριν για τα ελαστικά στα αυτοκίνητα. Ναι, είναι σαν να οδηγούμε ένα αυτοκίνητο με σκασμένο λάστιχο. Κάτι το οποίο βέβαια κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε ανισορροπίες και σε ατυχήματα. Τι εννοώ δηλαδή, ότι η Τραπεζική Ένωση φτιάχτηκε βασιζόμενη στην ε, προϋπόθεση της μακροοικονομικής ανάκαμψης, κάτι το οποίο όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, παρόλο που βελτιώνεται η κατάσταση. Και απόδειξη αυτού είναι ότι εξακολουθούμε να συζητάμε πώς θα αντιμετωπίσουμε διάφορες κρίσεις που έχουμε κληρονομήσει, ενώ δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία πια. Στο σημερινό πλαίσιο λοιπόν, οι σκληρές συνθήκες για κάθε πρόσβαση στα πλαίσια είτε των εθνικών κανόνων είτε της οδηγίας ανάκαμψης και εξυγίανσης τραπεζών ε, συγκεντρώνονται γύρω από το ότι χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο, ότι έχουμε ένα περιβάλλον χαμηλής απόδοσης, ε, υψηλά επίπεδα MPLs και όλα αυτά οδηγούν σε μεταφορά πλούτου και διακινδυνεύεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν οι εθνικές ανησυχίες και η ευθύνη ε, συζητιώνται σε εθνικό επίπεδο και διαθέτουν εθνικά εργαλεία, τα οποία όμως είναι όλο και πιο αποδυναμωμένα. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος καλός συντονισμός. Είπα και πριν ότι λείπουν κάποια στοιχεία. Ακόμα τώρα δεν έχουμε ένα κοινό δίκτυο ασφάλειας ούτε για τους καταθέτες, ούτε για, την, για το Ταμείο Εξυγίανσης. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά μέσα μείωσης του κινδύνου, δεν έχουμε όμως σχεδόν κανένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ τις προϋποθέσεις για την ε, προληπτική ανακεφαλοποίηση και πρέπει να δούμε πώς παρεμβαίνει το Ταμείο, το Ενίο Ταμείο Εξυγίανσης και τι γίνεται και με την εφαρμογή του MRL. Όταν μιλάμε για 5% τλάκα και 18% MRL, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί πολύ δύσκολα να λειτουργήσει το Ταμείο Εξυγένσης. Και αυτό είναι μεγάλη δυσκολία όταν θέλουμε να μιλάμε για σταθερότητα και να βασιζόμαστε στις τράπεζες που έχουν χάσει σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόλο που είχαν παλιά είτε επειδή οι ευθύνες τους έχουν να κάνουν περισσότερο με τις καταθέσεις είτε επειδή εξακολουθούν να χρησιμοποιούν στοιχεία κινδύνου. Για το MRL πιο συγκεκριμένα, ούτε και αυτό είναι χωρίς αδυναμίες. Δυστυχώς δεν λάβαμε υπόψη μας πλήρως το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας με τους στόχους τους που προβλέπονται από το MRL όταν αυτό αρχίσει να ισχύει. Που σημαίνει ότι οι τράπεζες που βασίζονται κυρίως σε καταθέσεις θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση για να εκδώσουν μέσα MRL ή θα μπορέσουν να το κάνουν με ιδιαίτερα υψηλό κόστος και με περιορισμό πρόσβασης στις αγορές. Πιστεύω ότι οι απώλειες είναι απώλειες που πρέπει να αναλαμβάνουν οι μέτοχοι, οι δύσμες να γίνεται διάσωση και όχι ο κόσμος και οι φορολογούμενοι και το δημόσιο. Γι' αυτό πρέπει να δούμε ποιος είναι επιλέξιμος για MRL και να φροντίσουμε να δώσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή για τελειώς πρέπει να ξέρουμε ότι επεκτείνουμε το MRL σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ το TLAC περιορίζεται μόνο στις, στους συστημικά σημαντικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Δεν θέλω βέβαια να ολοκληρώσω χωρίς να κάνω έκκληση για μια συστημική προσέγγιση MPL που να με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και να τα σκεφτούμε πολύ γιατί την σταθεροποίηση τη χρειαζόμαστε. Δεν είχε προβλεφθεί, αλλά τώρα χρειαζόμαστε πάρα πολύ τέτοια σταθεροποιητικά μέσα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλους σας και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε και να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν διαθέτει ακόμα και αυτό προς όφελος και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της διασφάλισης της δανειοδότησης αλλά και προστασίας των καταθετών. Και άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ και σίγουρα η συζήτηση αυτή είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Ευχαριστώ πολύ, Ελίζα. Ναι, όχι μόνο έχουμε σκασμένο ε, ε, λάστιχο, δεν έχουμε και αρκετέ ρόδε. Ελπίζουμε αυτή η δέσμη μέτρων ε, να δημιουργήσει κάποιε από αυτέ. Ευχαριστώ όλου του ομιλητέ. θα αναλάβει τώρα η Σουίνμπερν την Προεδρία. Θα επανέλθω σύντομα. Thank um, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε επαναδιαπραγματευτεί τον χρόνο ομιλία. Τρία λεπτά για τον κάθε ομιλητή γράφουν οι σημειώσει μου, ε, ενώ μου είπαν δύο. Θα δώσουμε τα τρία λεπτά όπω είχαμε πει αρχικά, αλλά αν μπορέσετε να περιορίσετε το χρόνο ομιλία σα, ε, θα είμαι πολύ ευγνώμων. Θα ακούσουμε πρώτα τις πολιτικές ομάδες. Εάν μας το επιτρέψει ο χρόνος μετά, ε, θα έχουμε και συζήτηση Catch the Eye. Έχουμε πρώτα τον Μπούρκα Πάλτς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές μας. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας ε, αναθεωρήσαμε τις κεφαλαϊκές απαιτήσει για τις τράπεζες κάτι που οδήγησε στη δημιουργία του Συμβουλίου ε, για τον ε, ενιαίο μηχανισμό ε, εξυγίανσης. Και έτσι καταφέραμε ο Ευρωπαίος φορολογούμενος να προστατεύεται σε περίπτωση αποτυχίας των τραπεζών. θα ήθελα να συμφωνήσουμε πάνω στο στόχο αυτόν. Ε, ήδη κατά την εφαρμογή των ισχυών των κανόνων ε, αναζητώνται παρεκκλήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω από τον κύριο Τέντε και την ε, αγαπητή μου φίλη την Ελίζα Φερέρα να μου απαντήσουν στο εξής όσον αφορά την αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τις ε, τράπεζες, πώς μπορούμε να φροντίσουμε να προστατεύεται καλύτερα ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, σε τι θα πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να διασφαλίσουμε ε, αρκετό MRL και δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τους κανόνες αντί να τους περιορίσουμε. Επίσης, όσον αφορά τις ε, εξαιρέσεις ε, του ΤΙΛΑΚ για τις ε, συστημικά σημαντικές τράπεζες, πώς το βλέπετε αυτό και πιστεύετε ότι αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί και στα πιστοτικά ιδρύματα που δεν είναι GCs, που δεν είναι συστημικά σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ, Μπουρκχαρτ. Περβάνς Περές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προσκεκλισμένους. Να επενθυμίσω ότι σε αυτό το πακέτο υπάρχει ένα κείμενο που δεν σήμερα επί τραπέζης, είναι η χρεοκοπία. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό για την ισορροπία, να το πούμε. Να αναφερθώ στο θέμα της ιεράσχησης των πιστωτών. Το ανέφεραν οι προσκεκλημένοι. Θέλω να επαληθεύσω μαζί τους σε ποιο βαθμό αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατεπηγόντως και αν οι όροι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της αναθεωρήσεως σε ξεχωριστή πρόταση απαιτεί επιταχυμένη εξέταση. Κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως σε αυτή τη φάση. Δεύτερον, η μείωση του κινδύνου. Περί τίνος πρόκειται. Έχω εντυπωσιαστεί από το επιτελεστέν έργων μέσω του πακέτου για τις τράπεζες, η μείωση του κινδύνου είναι η είσοδος στην προσέγγιση. Απευθύνομαι προς τους προσκεκλημένους. Θεωρώ ότι είναι πολύ ε, κοντόφθαλμη προσέγγιση αφορά τη μείωση του κινδύνου. Ο οικονομικός κίνδυνος συνολικά ε, γίνεται, γίνεται με, αντιληπτός με κακό τρόπο, με λαθασμένο τρόπο. Λοιπόν, Έχουμε μια νομοθεσία του σημαντικά χρησιμοτικά ιδρύματα που δεν λαμβάνει υπόψη τι εξωτερικές πτυχές κινδύνων, ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακος, χρήση του άνθρακα. Υποτιμούμε έναν οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κίνδυνο, αν υποτιμούμε αυτούς τους κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Εξετάζει τη βιώσιμη χρηματοδότηση μήπως να χρησιμοποιήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία για να συντονίσουμε το χρηματοδοτικό κανονισμό και τις ρυθμίσεις με τους στόχους μειώσεως των κινδύνων από πλευράς κλίματος ή από πλευράς ενεργείας. Μήπως πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα πράσινα και καστανά στοιχεία ενεργητικού green and brown assets που είναι στους πυλώνες 1 και 2 ή πυλώνες 2 και 3 ή αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στο επίπεδο της ομάδας βασιλείας. Το θέμα της αναλογικότητας αναφέρθηκε εκτενώς. Εξού και ερώτησή μου. Μήπως πρέπει να, πρέπει να έχουμε ορισμό της αναλογικότητας αυτής. Πρέπει να αναρμονίσουμε τις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο CRD και στο CRR και αυτή την νέα της αναλογικότητας να διαθρώσουμε γύρω από τρεις έννοιες. Μέγεθος, περίπλοκος χαρακτήρας, περιπλοκότητα και ύπαρξη επίπεδου κινδύνου ε, ορίζοντας ε, ποιος ακριβώς κίνδυνος είναι αυτός που θα πρέπει να την υπόψη. Ευχαριστούμε. Περβάς. Άργησε ο συνάδελφος από το ECR γιατί είναι σε ψηφοφορία. Θα σας διαβάσω εγώ την ερώτησή του που έχει να κάνει με τα μέσα του μορατόριου στο 10α. Υπάρχουν δύο είδη που προτείνονται. Το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την εξυγίανση που μέχρι πέντε μέρες έχει στη διάθεσή του οργανισμό για να τα αποκριθεί και η δεύτερη περίπτωση είναι όταν έχει ήδη αρχίσει η εξυγίανση οπότε οι αρχές πρέπει να εκτιμήσουν το ενεργητικό για να δούνε ποια θα είναι η διαδικασία εξυγίανσης που θα ακολουθήσουν. Ο Σκιώδης από το ECR έχει κάποιες αμφιβολίες αυτή την διακοπή για πέντε μέρες πριν μπει σε εξυγίανση τράπεζα θεωρεί ότι είναι υπερβολικά πολλές, ότι υπάρξει στρέβλωση, ότι εμποδίζεται συνεργασία και θεωρεί ότι τότε θα οδηγηθεί όντως σε ο οργανισμός. Σε πέντε μέρες από την άλλη μεριά να υπάρξει εκτίμηση του ενεργητικού είναι πολύ λίγο. Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες, μπορεί να χρειαστούν έξι μήνες. Η σημερινή οδηγία BRRD προβλέπει τις πέντε μέρες. Όμως επειδή πρόκειται για μια ελάχιστη εναρμόνιση, μπορούν να επεκτείνουν τις εθνικές αρμοδιότητες οι χώρες μέλη και αν χρειαστεί να εφαρμόσουν και άλλα μορατόρια. Το ECR θα ήθελε να ακούσει λοιπόν από το πάνελ κατά πόσο πιστεύουν ότι αυτές οι νέες εξουσίες μορατόριου είναι χρήσιμες ή όχι. Κατά πόσο θα βοηθήσουν σε περιπτώσεις στρες και μήπω πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενη ερώτηση, λέει και κλείνει το μικρόφωνο τη ομιλητής, δεν ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Το πακέτο αυτό, και καλημέρα Ελίζα, προσπαθεί να αποφύγει μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε να κοιτάμε και προς το μέλλον. Και δικιά μου πεποίθηση είναι ότι τελικά ε, όταν μιλάμε για τις τράπεζες δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Διότι υπάρχει το software και οι ψηφιακές ικανότητες. Αν δεν κοιτάξουμε λοιπόν το λογισμικό, το software, βλέπω εγώ πρόβλημα, γιατί για οργανισμούς που είναι στην Ευρώπη τότε πρόκειται για ένα ενεργητικό το software. Πρέπει δηλαδή να αφαιρεθεί από το Tier 1, από την πρώτη κατηγορία. Και επίσης αυτό χρησιμεύει και ως κίνητρο ή αντικίνητρο για επενδύσεις στην καινοτομία και μπορεί να οδηγήσει και σε θέμητο ανταγωνισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, καταγράφεται σαν άλλο κεφάλαιο και πρέπει να αφαιρεθεί. Και αν το συγκρίνουμε με την ε, ε, ευρωπαϊκή κατάσταση υπάρχει το άλλο ενεργητικό που επίσης ε, παίζει ρόλο εδώ. Οπότε δεν συμφωνείτε ότι οι επενδύσεις σε software θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τον κλάδο. Και επιπλέον, αν κοιτάξουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συστήματα ισοτιμίας, τότε κεφαλαϊκά καθεστώτα από άλλες χώρες που δεν προβλέπουν την αφαίρεση του software δεν λαμβάνονται υπόψη ως διάκριση. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι κάτι που δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό τελικά. Και τέλος η ερώτησή μου, με που έχω χρόνο, έχει να κάνει με τις ψηφιακές ικανότητες γιατί στους καιρούς αυτούς fintech ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο στον οικονομικό τομέα. Όλοι αγωνιζόμαστε και καταλαβαίνετε ποια είναι η ερώτησή μου. Έχει να κάνει με την καινοτομία. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι δημιουργεί μειονέκτημα για το τραπεζικό τομέα προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί όλους τους άλλους τους κλάδους κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους πράσινους, παρακαλώ. Καλημέρα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ε, δηλώσω τις αρχές μας. Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να είναι δημόσιες. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις τράπεζες θα πρέπει να ε, είναι του δημοσίου τομέα. Έχουμε λοιπόν επιφυλάξεις όσον αφορά όλους αυτούς τους κανόνες, διότι δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να ρυθμίσει κανείς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, διότι είδαμε πώς απέτυχαν οι ρυθμίσεις του παρελθόντος. Τούτου λεχθέντος, έχουμε μια σειρά νομοθετικών στοιχείων ιδιαίτερα περίπλοκων και αμφιβάλλουμε ότι θα συμβάλλουν ε, στην αντιμετώπιση του προβλήματος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι υπερβολικά μεγάλα για να μπορούμε να τα αφήσουμε να χρεοκοπήσουν. Διασφαλίζουμε στους ε, εργαζόμενους, στους ανθρώπους, ότι δεν ε, θα υπάρξει άλλος επιμερισμός των απολειών των τραπεζών στους φορολογούμενους. Και πολύ συγκεκριμένα έχω μία παρατήρηση για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης απολειών, TILAC. Το ποσοστό, μάλλον, ε, ναι, το ποσοστό θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να αυξηθεί από τη Γερμανική Τράπεζα. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις και των ε, άλλων ομιλητών το TILAC θα εφαρμοστεί σε 13 τράπεζε εδώ στην Ευρώπη και εγώ αναρωτιέμαι για τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επίση είναι συστημική σημασία. Δεν θα πρέπει να πληρούν τι ίδιε απαιτήσει ή να υπάρχουν τουλάχιστον κάποια προληπτικά μέτρα. Όσον αφορά την προληπτική ανακεφαλοποίηση, αυτή εφαρμόστηκε στην Ιταλία. Δεν δείχνει την ανικανότητα του συστήματος να αντιμετωπίσει απώλειες και ιδιαίτερα τα κακής ποιότητας ε, δάνεια στο τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η αρχή που θα εφαρμόσουμε στο μέλλον. Αυτό ουσιαστικά οδηγεί στο να υπομειστεί ο φορολογούμενος ε, της απώλειας των τραπεζών. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με το ποσοστό μόχλευσης και τον καθορισμό του συμπεριλαμβάνονται διάφορα περιουσιακά στοιχεία διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και θα ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις των ομιλητών μας ε, πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα ιδιαίτερα να απευθυνθώ στον κύριο Ραποριά, ελπίζω να προφέρω σωστά τα όνομά σας. θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για την νέα κατηγορία τους, ε, ε, τους σημαντικούς μη προτιμησιακούς πιστωτές. Ευχαριστώ κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς χαίρομαι που σε βλέπω ξανά εδώ Ελίζα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Και μια ερώτηση για σένα. Εργαστήκαμε μαζί και πάντα υποστηρίζαμε διπλή στρατηγική. Να μειώσουμε τους κινδύνους και να υπάρχει και επιμερισμός των κινδύνων. Μέχρι τώρα έλεγε ότι ο επιμερισμός των κινδύνων δεν λειτουργεί σωστά. Πώς το βλέπεις εσύ. Τι θα πρέπει να προτείνει το Κοινοβούλιο για να ενισχύσει το κομμάτι για τον μερισμό του κινδύνου της Τραπεζικής Ένωσης. που στην κυρία Νουή τώρα. Ευχαριστώ για την άποψή σας και για τις προτάσεις σας. Ζητάτε περισσότερη Ευρώπη στο πακέτο. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τα περισσότερα από αυτά που είπατε. Άρα, μία ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση αυτό που δεν αναφέρατε ήταν στη μακροοικονομική εποπτεία και τα εποπτικά εργαλεία. Μπορείτε να δώσετε στο Κοινοβούλιο συγκεκριμένες προτάσει σχετικά με αυτά. Δεύτερη ερώτηση. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής δυστυχώς κατέφθασε χωρίς ε, μια ποσοτική αξιολόγηση συνεπειών. Δεν ξέρουμε αν μειώνεται πράγματι ο κίνδυνος ή όχι. Οι αλλαγές του πυλώνα 2 και των κατευθυντηρίων γραμμών αυτού, ούτω ώστε κεφαλικές απαιτήσει να μετατραπούν σε κεφαλαιοκικούς προσανατολισμούς για το SSM, έχει αποτέλεσμα 155 δισεκατομμύρια ευρώ μετατροπής από πρώτες δεσμευτικές απαιτήσει σε κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό σημαίνει ίσως ότι δεν είναι πακέτο περιμειώσεως κινδύνων, αλλά εμπεριέχεται και ένα αποτέλεσμα αυξήσεως κινδύνου. Εξού και ερώτησή μου. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να ποσοτικοποιήσουμε τα αποτελέσματα για το ΣΕΣΕΜ των διαφόρων μέτρων που προτείνονται στο πακέτο. Τέλος. Απευθυνόμαστε στον κύριο Ανδρέα Ένρια και σε εσά κυρία Νουή. Ε, το ECB και το EBA ε, μπορούν να κάνουν προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πώς να ενισχύσουν την ε, αναλογικότητα στους κανονισμούς περί τραπεζών ακούγονται πολλές επικρίσεις που είναι επιβλαβείς για τις φήμες των μικρών χρηματοστικών ιδρυμάτων. Θα ήταν καλό αν τα δικά σας θεσμικά όργανα μπορούσαν να υποβάλουν προτάσεις για μας, τους νομοθέτες, για να ενισχύσουμε την αλογικότητα. Τι ούτω τρόπος αυξάνοντας την υποστήριξη για την Τραπεζική Ένωση, για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Ευχαριστούμε. ΙΕΝΕΦ. Μπαινό. Α, ή όχι. Βάλε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομε. Η πρώτη απευθύνεται προς τον κύριο Λαμποριέ, κύριο Λαμποριέ και αφορά το θέμα της διαφάνειας. Συζητούμε με τους άλλους και όδης εισηγητές το θέμα αυτό για την αναθεώρηση της οδηγίας BRD. Και ένα από τα προβλήματα που τίθεται είναι της διαφοροποίησης των αποφάσεων του Single Resolution Board σε κάποιες περιπτώσεις. Και το να τεθεί ε, σε σε μια τράπεζα μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει συστημική σημασία. Και είναι ευαίσθητε οι πληροφορίε που πρέπει να χορηγηθούν. Άρα κάποιε πληροφορίε πρέπει να παραμείνουν κρυφές από το κοινό για να μην δημιουργηθεί πανικό στην αγορά. Διαρωτώ με, μπορεί να υπάρχει περίοδος χρονική μετά από την οποία δεν είναι πλέον ευαίσθητες πληροφορίες. Συνεπώς μπορούν να δημοσιευθούν οι λόγοι για τη λήψη αποφάσεως, να επικρατήσει διαφάνεια. Μπορούμε να καθορίσουμε κάτι τέτοιο, μια χρονική περίοδο μετά την οποία μπορεί να επικρατήσει διαφάνεια και να εμφανίζονται οι λόγοι για τη λήψη μιας αποφάσεως δεν ξέρω, έξι μήνες, ένα χρόνο, για να δώσουμε κίνητρο για εφαρμογή ορθής πρακτικής, όπως θα ήταν η διαφάνεια στον αφορά τις αποφάσεις. Μετά μια άλλη ερώτηση. Όλοι γνωρίζουμε καλά πώς ενδιαφέρονται οι κερδοσκόποι για την αγορά των non-performing loans, των κόκκινων δανείων. Το είδαμε από τη διαχείριση που ήδη έλαβε χώρα κάποιων περιστάσεων στην κρίση που οδήγησαν στην πώληση κάποιων πακέτων αυτών των δανείων. Επολύθησαν σε χαμηλότατες τιμές. Και μετά, όταν αγοράστηκαν, αγοράστηκαν στις τιμές πολύ ψηλότερες. μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας, πώς γίνεται η διαχείριση των κόκκινων δανείων ούτως ώστε να μην θεωρούν οι κερδοσκόποι ότι είναι μια πανεύκολη αγορά για αυτούς και πολύ αποδοτική. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν και τη χρήση δημοσίων πόρων. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν οι κερδοσκόποι να ενδιαφερθούν πολύ όσον αφορά τη διαχείριση των ε, κόκκινων δανείων. Thank you for Ευχαριστούμε. ΕΝΕΦ. Όχι. Α, ωραία. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις και κάποιες πολύ ειδικέ. Δύο-τρία λεπτά ο κάθε προσκεκλημένος μας παρακαλώ για να απαντήσει. Αν δεν θέλετε, δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Το αφήνουμε σε εσά. Ποιος θα αρχίσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όντως, κάποιες δεν θα μπορέσω να απαντήσω. Αλλά θα αρχίσω με το εξή για την προστασία του φορολογούμενου, τις ε, προληπτικές κεφαλοποίησεις και την απόδοση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το στοιχείο κλειδί εδώ είναι ότι μπορεί να έχετε περιπτώσεις όπου η τράπεζα ή οι τράπεζες δεν είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν, αλλά να έχουν έναν ισολογισμό γεμάτο με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οπότε η απόδοση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Συνεπώς έχουν ως τράπεζες πολύ χαμηλή απόδοση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε υπάρχει η δυσκολία να δοθεί και κρατική βοήθεια ώστε να προχωρήσει η τράπεζα. Όμως το στοιχείο κλειδί εδώ είναι ότι πρέπει να γίνει κάτω από τα πολύ αυστηρά κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγένση και να αφροντίσετε η τιμή ε, για το ενεργητικό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέω ότι τη χρήση του μηχανισμού αυτού δεν πρέπει να το θεωρήσουμε ως απόκληση από την BRRD, αλλά είναι μια συγκεκριμένη χρήση της οδηγίας αυτής κάτω από πολύ δικές συνθήκες. Και για το τελευταίο που ακούσαμε, στην περίπτωση αυτή έχετε 12-15 αγοραστές, ενώ οι, που είναι πολύ συγκεκριμένοι, ενώ οι πολιτές είναι πολύ διασκορπισμένοι. Οπότε πρέπει να υπάρξει αυτή η αντιστοιχία για να πετύχουμε μια καλύτερη τιμή και να είναι η αγορά πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Όσον αφορά τώρα την ιεραρχία των πιστωτών. Εμείς στηρίζουμε τις προτάσεις και θυμάμαι ότι και το προσωπικό της CBA αυτό ακριβώς πρότεινε την εποχή δηλαδή που ετοιμάζαμε την οδηγία για την ανάκαμψη και για την εξυγίανση. Οπότε μας ικανοποιεί η πρόταση και πιστεύουμε ότι επειδή είναι ιδιαίτερα ρευστές οι αγορές, οι τράπεζες θα πρέπει να επιταχύνουν τη συμμόρφωση προς την δομή του παθητικού τους και πρέπει και νομοθετικά να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Για την αναλογικότητα, ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά ζητήματα εδώ. Το ένα είναι ότι έχουμε ήδη πολλή αναλογικότητα στο σύστημα. Σήμερα μια μικρή τράπεζα συμμορφώνεται 10% με το δικό μας πλαίσιο αναφοράς. Μερικές φορές είναι δύσκολο γιατί το πακέτο έχει υψηλέ προδιαγραφές, οπότε ευτυχώς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις για, πώς να το πω, ένα ψηφιακό εγχειρίδιο κατά κάποιο τρόπο που επιτρέπει στις τράπεζες να καταλάβουν με τι ακριβώς πρέπει να συμμορφώνονται. Αυτό θα το αναπτύξουν περισσότερο και ευχαριστούμε για την πρόταση. Το δεύτερο στοιχείο είναι η απλοποίηση του βάρους της συμμόρφωσης, κυρίως στον τομέα της αναφοράς και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να βοηθήσουμε. Και τα διάφορα επιπλέον στρώματα ε, που μπαίνουν στην αναφορά πρέπει να διευκρινιστούν. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχουν ακριβώ κάποια τέτοια στρώματα όπου οι απαιτήσει δεν ανταποκρίνονται ε, στις περιπτώσεις των μικρών τραπεζών. Πρέπει λοιπόν να μειωθούν. Όσον αφορά τώρα το TILAC, εμείς το επενθύμησε και ο Ντομινίκ, θελήσαμε να επεκτείνουμε τις απαιτήσει αυτές και σε άλλα, άλλους οργανισμούς συστημικά σημαντικούς Οπότε συμφωνούμε με μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά το τηλεκτρονική ικανότητα απορρόφησης απολειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ε, κυρία Νουή. Ευχαριστώ. Τι είναι η προστασία του φορολογούμενου. Δεν γνωρίζουν ε, οι μικρές ε, τράπεζες ότι μπορεί να υπάρχει, μάλλον μικροί επενδυτέ, ότι μπορεί να χάσουν επειδή ακριβώς θα υπάρξει bail-in όταν επενδύουν σε μικρές τράπεζες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τεχνικές, αλλά θα υπάρξει δημοσίευση ενός ε, μεγαλύτερου κειμένου Υπάρχει ήδη μια εισαγωγή, αυτός που έκανε την ερώτηση δεν έχει παρά να πάει στο site να το δει. Τώρα όσον αφορά τι μειώσει από το ILO τμήμα, πρέπει να υπάρξει απορρόφηση των απολειών, όπως είπαμε, και εδώ υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία επιτρέψαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όσον αφορά τις ILS equities. Τώρα, υπάρχει μια μείωση των εξαιρέσεων. Θα ισχύσει από το 2019. Η αξία του IT δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην ε, απορρόφηση απώλειας. Πάντως, για το ότι οι πληροφορίες πρέπει να είναι Δηλαδή, δίνονται στο κοινό, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να κάνουμε εποπτεία αν συγκεντρώνουμε τους προβολείς σε κάθε δραστηριότητα. Τότε θα υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος παράοφελος. Και όσον αφορά το TILAC, τη συνολική ικανότητα απορρόφηση απολειών και τι σημαίνει για τι τράπεζε, στην Ευρώπη έχουμε το MRL, την ελάχιστε απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτέ υποχρεώσει. Σίγουρα χρειάζεται μια αναλογικότητα γιατί οι μικρέ τράπεζε είναι λιγότερο συστημικά σημαντικέ στην αγορά. Τώρα για την αναλογία μόχλευση. Πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στον ορισμό που ακολούθησε η Βασιλεία. Οποιαδήποτε εξαίρεση μειώνει την αξία αυτού του μέσου και τη διαφανεία. Αν χρειάζεται εξαίρεση για κάποια κατηγορία τραπεζών, τις ε, αναπτυξιακές τράπεζες για παράδειγμα, αυτό θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, να υπάρξει ένα χαμηλότερο ποσοστό μόχλευσης για αυτές, αλλά να είναι γνωστό ό,τι παρεκκλήσεις υπάρχουν, να υπάρχουν με διαφάνεια. Αν υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη μακροοικονομική ε, ενημέρωση, εναρμόνιση όσον αφορά την ε, μακροπροληπτική εποπτεία, ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να πετύχουμε περισσότερη εναρμόνιση Άλλη ερώτηση για τις απαιτήσει του πυλώνα 2 όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές. Κάνει υπάρχει ενίσχυση κινδύνου. Δεν θα έλεγα, απλώς καθυστερεί η στιγμή που θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος, γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές ζητούν να συγκεντρώσουμε διάφορα στοιχεία και όταν έχουμε συζητήσει και έχουμε αναλύσει με τον κεφαλαικό σχεδιασμό με την τράπεζα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλα μέτρα. Οπότε, ναι, μεν υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά ε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής στην οποία οφείλεται η καθυστέρηση, μειώνεται, πιστεύω, ο κίνδυνος. Αναλογικότητα, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει μέσω της συχνότητας, αλλά μέσω της ακρίβειας της ε, του πρότυπο αναφοράς. Ζητούμε από τις ε, τράπεζες να έχουν ήδη έτοιμο το πληροφορικό τους σύστημα. είναι ισοδική σημασία για μας για να προβούμε σε εποπτεία, να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για την τράπεζα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό πιο γρήγορα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, είναι αλήθεια, να εισάγουμε δηλαδή το στοιχείο της ακρίβειας στις αναφορές που απαιτούμε. Τώρα τις ε, φτηνές τιμές για τα MPLs. Όταν έχουμε μη εξυπηρετούμενη έκθεση στην αγορά, ε, τότε οι πολιτές δεν έχουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών Γι' αυτό και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής έχει πολλά πλεονεκτήματα. Δεν σημαίνει αλληλεγγύη στη χρηματοδότηση στην κάλυψη των απολειών, απλώς προσφέρει περισσότερη διαπραγματευτική ικανότητα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πάντως να βελτιώσουμε το νομικό πλαίσιο στις χώρες μέλη. εξοδικαστικές μέθοδοι ε, κάλυψης. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την κάλυψη των ε, μη δημοσίων εγγύσεων. Θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι ήδη μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λάβει διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την ιεράρχηση των πιστωτών, την ξεχωριστή αυτή πρόταση και όπως είπε ο Ανδρέα, την πρόταση αυτή την θεωρούμε ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δέσμη μέτρων, με την έννοια ότι απέχει από τις τροποποίησεις που προτείνονται στην υπόλοιπη δέσμη μέτρων, διότι εισάγει ένα επιπλέον επίπεδο ε, σε περίπτωση που έχουμε κρίση ή που έχουμε ε, διάλυση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το επιπλέον επίπεδο, διότι αυτό θα δώσει ασφάλεια στους επενδυτές, θα βελτιώσει το επίπεδο MRL e και γι' αυτό ε, στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν και μάλιστα όσο πιο γρήγορα εφαρμοστούν αυτά τόσο το καλύτερο χωρίς, ε, με την επιφύλαξη μάλλον των προτάσεων που ήδη εφαρμόζονται. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εφαρμοστούν και αυτοί οι κανόνες όσο γίνεται πιο γρήγορα για να αποφύγουμε την καθυστέρηση. Όσον αφορά το μορατόριο. Ναι, η πρόταση αυτή αποτελείται από δύο ξεχωριστά ε, στοιχεία και εάν συνδυάσουμε τα δύο αυτά στοιχεία με το τρίτο που ήδη υπάρχει, θα μπορούσαμε να έχουμε Ε, μεγαλύτερες δυνατότητες και είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις. Δεν είναι δυνατόν ε, να ανασταλούν όλες οι δραστηριότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όσον αφορά τα δύο moratorium, υπάρχει το ερώτημα τι γίνεται εάν έχουμε και ένα δεύτερο. Θα υπάρξει διακοπή ανάμεσα στα δύο αυτά στάδια ή όχι και όπως υπόθηκε σίγουρα είμαστε υπέρ του μορατόριου διότι έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο για την εφαρμογή των μέτρων. Εάν έχουμε δύο μορατόριου θα πρέπει να γίνει στενός συντονισμός ε, ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Υπάρχουν και άλλα θέματα πέρα από τις καθυστερήσεις. Το θέμα του πεδίου εφαρμογή ε, είναι ζωτικής σημασίας. Αν ε, δεν έχουμε ε, αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογή όσον αφορά την ευθύνη, θα είναι και περιορισμένη η προστιθέμενη αξία του μορατόριου. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και όπως είπα και εγώ κατά την εισαγωγή μας, κατά την εισαγωγή μου, Είμαστε υπέρ του οι τράπεζες να έχουν επαρκές χρέος για τη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάσωσή τους. Όλες οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να δημιουργήσουν αυτό το επιπλέον επίπεδο το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε την ευελιξία για να τροποποιήσουμε την προσέγγιση χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς. Μάλιστα, όσον αφορά την ποιότητα, το θέμα αυτό και την ιεράρχηση των χρεών, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και ίσως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ποιότητα με αρκετά μικρό τίμημα. Και τέλος, όσον αφορά το θέμα της διαφάνειας, όπως υπόθηκε ήδη, από την πλευρά της εξυγίανσης αντιμετωπίζουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα και θα πρέπει να ε, γίνει διάκριση ανάμεσα στην ε, περίοδο σχεδιασμού και στην περίοδο ε, εφαρμογής της εξυγίανσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά θα πρέπει να γίνει προσεκτικά αυτός ο σχεδιασμός της εξυγίανσης. Δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή η ιδέα να κοινοποιείται αμέσως ο στόχος. Ε, σημαντικό είναι οι τράπεζες να γνωρίζουν ότι θα πρέπει ε, σε βάθος χρόνου και βήμα-βήμα να δημιουργήσουν αυτό το επιπλέον επίπεδο για το MREL. Θα πρέπει να εξεταστούν τα στοιχεία του παθητικού και το, η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ θετική όσον αφορά την πτυχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θα σχολιάσω εγώ ένα-δύο θέματα που μας αφορούν όσον αφορά την έκθεση την green and uh, brown exposures, τις εκθέσεις αυτές, θα πρέπει αυτά να καλύπτονται το πλαίσιο που θέσαμε. Ε, εξετάσαμε την έκθεση την πιστοτική σε διάφορες τράπεζες για να δούμε αν λάβαναν υπόψη ότι επίσης έπρεπε να λάβουν υπόψη κλιματολογικούς κινδύνους στην έκθεσή τους και η εμπειρία μας ήταν ότι εν γέννη το κάνουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Κάποιοι κινδύνοι είναι πάρα πολύ μακροπρόθεσμοι και ο κίνδυνο είναι να ακολουθείτε πολύ βραχυπρόθεσμη προσέγγιση. Δεν είμαι πεπισμένο ότι χρειαζόμαστε έναν κάποιον κανονισμό. Χρειαζόμαστε όμως να δοθεί κάποια προσοχή από τι ρυθμιστικέ αρχές. Όσον αφορά ψηφιακέ δεξιότητε και αμοιβέ, αυτό ε, είναι πολύ επίκαιρο για τη Σουηδία, γιατί όπως ε, είναι πολύ μεγάλο ο τομέα στη Σουηδία. Ε, δεν νομίζω ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν ανθρώπους από την, από την FinTech ε, με περιορισμού όσον αφορά τι αμοιβέ που θα προβλέπονται από τον κανονισμό περί τραπεζών. Νομίζω ότι δύσκολο να, να αλλάξει νοοτροπία σε μια τράπεζα. Όταν κάποιοι καινοτομούν να προσλαμβάνονται από τράπεζα δεν είναι πρόβλημα. Οι τράπεζες πληρώνουν πολλά περισσότερα χρήματα από ό,τι εμείς. Το άλλο που ετέθη για τα εσωτερικά μοντέλα και τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην λαμβάνονται υπόψη συστημική κίνδυνη. Τα εσωτερικά μας μοντέλα για τα κίνητα είναι περίπου ο κίνδυνος στα 5%. Δεν έχουν απώλειες πιστώσεων όσον αφορά τη στέγαση στη Σουηδία. Για λόγους νομικούς και κοινωνικούς ε, λόγω του συστήματος που έχουμε, προνοίας. 5% είναι, είναι πολύ χαμηλή έκθεση. Οπότε θα προσθέσουμε κεφαλαιοχική απέτηση στον πυλώνα 2 λόγω συστημικών κινδύνων. Ίσως αυτό να είναι ένα φύκτο όμως και περιορισμένο στο τραπεζικό πακέτο, άρα χρειάζεται ευελιξία. Τέλος, ποσοστό μόχλευσης μας ικανοποιεί. Πρέπει όμως να είναι χαμηλότερο από τον σταθμισμένο κίνδυνο, από το κεφάλαιο που απαιτείται βάσει σταθμισμένου κινδύνου. Αλλιώς μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο. Το ποστό μόχλευσης συνεπάγεται το ίδιο κεφαλουχικό, α, κεφαλουχική απέτηση για στοιχεία ενεργητικού με κίνδυνο όπως και για στοιχεία ενεργητικού ανευκίνδυνου. Οπότε το ποσοστό μόχλευσης δεν πρέπει να είναι κάτι δεσμευτικό, σαν μια φετηρία. Διότι εμποδίζει ε, τη διαμόρφωση τη σωστή των εσωτερικών μοντέλων. Ευχαριστώ. Η Ελίζα Φερέρα. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να καλύψω διάφορες ερωτήσεις. Το βασικό είναι το διαφορετικό επίπεδο και παρουσία των MPL σε όλο το σύστημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα βέβαια με την ίδια διάσταση παντού. Μην ξεχνάμε ότι κάποιες ε, ε, δικαιοδοσίες δεν έχουν τα NPLs που απορρέουν από συστημικές λύσεις που ελήφθησαν πριν από το 2013 στις δικαιοδοσίες αυτές, στις χώρες αυτές. Άρα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα μέσα στην ίδια χώρα. Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες ε, καθαρίστηκαν κατά κάποιο τρόπο πριν από το 2013 και πριν από την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγένση, ενώ αλλού παγιδεύτηκαν ε, τελικά και δεν υπάρχει λύση. Οπότε, οι απαιτήσει για επιπλέον καθάρισμα αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Και αυτό δημιουργεί και όρους που δεν είναι τελικά ισότιμοι για όλους και αυτό οδηγεί σε μεγάλη μείωση της αποδοτικότητας των τραπεζών. Το δεύτερο στοιχείο είναι το MRL. Αν θέλετε να διασώσετε μια τράπεζα, φυσικά και πρέπει να υπάρχουν ίδια μέσα για να γίνει αυτό. Όμως αν η απόδοση της τράπεζας στην ίδια περίοδο είναι πάρα πολύ χαμηλή και έχετε υψηλό επίπεδο NPL στον ισολογισμό, τότε το αίτημα για επιπλέον κεφάλαιο θα κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και θα υπάρξει τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών που μπορούν να πληρώσουν και των τραπεζών που που δεν θα μπορούν να πληρώσουν γιατί έχουν ε, προετοιμαστεί με ίδιους πόρους. Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό και η αναλογικότητα και η μεταβατική περίοδο είναι πράγματα που είναι ευπρόσδεκτα. Κάτι το οποίο είπε και ο Ντομινίκ πριν. Στο ζωτικό ζήτημα του Σβέν. Σβέν, ναι, και εγώ πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και πάλι μαζί σας. Πάντως, από πλευράς πακέτου Τραπεζικής Ένωσης δεν υπάρχει επιμερισμός κινδύνου, υπάρχει έλεγχος κινδύνου. Ο επιμερισμός είναι σε επίπεδο εποπτικού ελέγχου, σε επίπεδο εξυγένσης, αλλιώς δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει μηχανισμός για σταθεροποίηση. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο προς το παρόν. Κυρίως επειδή οι πιο σημαντικές συστημικά τράπεζες είναι αυτές που βλέπουν σαν πιο σταθερές, πιο παραδοσιακές οι καταναλωτές και άρα λιγότερο επικίνδυνες. Οπότε αν δεν καλύπτονται από ειδικά καθεστώτα κάποιες τέτοιες τράπεζες, τότε αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να πρέπει να διασωθούν οι μέσεις με καταθέσεις ή ακόμα και παλιό χρέος, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται για αυτό το σκοπό. Νομίζω ότι είναι ο χειρότερος τρόπος να πετύχουμε τον στόχο που αναφέρθηκε και να προστατεύσουμε τους φορολογούμενους. Γιατί τότε πρέπει να βρούμε διάφορα εναλλακτικά μέσα. Έχουμε παρατηρήσει τι έχει γίνει μερικές φορές με αυτά που τελικά δεν καταφέρουν να σταθεροποιήσουν το σύστημα, γιατί αυτό που γίνεται, γίνεται διάσωση και από καταθέτες και επενδυτέ που δεν έχουν πληρώσει για τη διάσωση μέση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η διάσωση. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε το πακέτο βέβαια, αλλά όλα μαζί, οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι νέοι κανόνες από τα 15, η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση, η εποπτεία για περισσότερο κεφάλαιο απαιτήσει και οι άλλες απαιτήσει για την έκδοση τίτλων που να μπορούν να διασωθούν οι δύο όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση που μας κάνει να πιστεύουμε ότι χρειάζεται συντονισμός και να αφήσουμε έναν χώρο να αναπνεύσει το σύστημα μέχρι την εφαρμογή όλων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που μόλις πήραν το λόγο. επέτρεψα τις ερωτήσεις για να ακούσουμε τις απαντήσεις και ζητώ συγγνώμη που δεν θα ακολουθήσουμε τώρα την ε, διαδικασία Catch the Eye, διότι μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Θα προχωρήσουμε τώρα ε, στην επόμενη σειρά ομιλητών μας. Ε, θα ακούσουμε την πλευρά των ενδιαφερομένων. Ζητώ συγγνώμη των προτέρων για την προφορά των ονομάτων. Καλό λοιπόν τον κύριο Κάρλ Πίτερ Σάκμαν Φάλης από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών. Πέντε λεπτά ο κάθε ομιλητής. Ε, παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις μας ε, για ε, τη νέα δέσμη μέτρων για το CRR, το CRD, το BRRD και το SRMR. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η δέσμη μέτρων, διότι χρειαζόμαστε μία, ένα διάλειμμα στην νομοθεσία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της νομοθεσίας προτού υποβληθούν νέες προτάσεις. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί τέλος στις νέες νομοθετικές προτάσεις ε, ε, για ένα διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σημαντικές και αποτελεσματικές ε, τροποποιήσεις ε, όσον αφορά το ποσοστό μόχλευσης ε, και αυτό είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις χρηματοπιστωτικές. Δεν είναι όμως απαραίτητο να γίνει πιο πολύπλοκη η νομοθεσία. Αυτό έχει να κάνει με τις εμπορικές και μη εμπορικές θέσεις στο CRR2, ε, το οποίο σημαίνει αυξημένη γραφειοκρατία για πολλές επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις ε, να μην τιμωρούνται ε, λόγω του εμπορικού χαρτοφυλακίου. Έχουμε άλλωστε τον κίνδυνο των τιμών της αγοράς και έτσι περνώ στις μικρές τράπεζες με πολύ περιορισμένο κίνδυνο, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη η εφαρμογή των προτάσεων θα πρέπει να οδηγήσουν σε αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο συνομοθέτης ε, με τη Βασιλεία 3 έχει εξισώσει τις ρυθμίσεις για 8.000 τράπεζες της Ευρώπης. Αυτό όμως το one size fits all, ε, το να έχουμε ε, τις ίδιες ε, ρυθμίσεις για όλες ε, τις τράπεζες, αυτό ε, δεν είναι καλή λύση. για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επηρεάζονται από αυτήν τη ρύθμιση. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της γραφειοκρατίας και ιδιαίτερα οι μικρές τράπεζες με πολύ περιορισμένο κίνδυνο επιβαρύνονται δυσανάλογα και αυτό το αυξημένο γραφειοκρατικό άχθος ε, αποτελεί επιχειρησιακό κίνδυνο για αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με περιορισμένο κίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες. Ε, κάποια μικρά στοιχεία αναλογικότητας δεν αρκούν ε, για τον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης. Προτείνουμε λοιπόν όλα τα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι μικρά και ε, με περιορισμένο κίνδυνο να απελευθερωθούν από αυτές τις υποχρεώσεις. Όλες δηλαδή οι μη συστημικές τράπεζες ε, να εξαιρεθούν από το άχθος αυτό. Και θα ήθελα να τονίσω ε, εδώ ότι μιλάμε για τις διοικητικές υποχρεώσεις όχι τις άλλες. Οι κανόνες της Βασιλείας προβλέπονται για μεγάλες τράπεζες. Δεν μπορούν λοιπόν να εφαρμοστούν στις μικρές τράπεζες ένα προς ένα. Θα θέλαμε περισσότερη αναλογικότητα όσον αφορά την εκαθάριση, τις ε, κοινοποιήσεις ε, και τα σχετικά τεστ. Κύριε Πρόεδρε, αναλυτικά Πολύ ευχαρίστως θα απαντήσω σε ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών μετά. Ε, ανέφερα αυτή τη στιγμή μόνο τα βασικά σημεία. Εάν εφαρμοστεί αυτή η αναλογικότητα στην Ευρώπη, θα είναι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανταγωνιστικά. στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης και του BRD Υπάρχουν υποχρεώσεις για τις ε, τράπεζες. Ε, δεν ε, είναι απαραίτητες όμως οι υποχρεώσεις σχετικά με το TILAC και το MREL για τις μικρές τράπεζες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φρεντερίκου Ντεά, επόμενος ομιλητής. επικεφαλής Σοσιατέ Ζωνεγάλ και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών. Καλώ ήρθατε κύριε Οντεά, έχετε το λόγο. Αγαπητέ Προέδρε, κύριε Γκαλτιέρη, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς να τονίσω ότι ομιλώ σήμερα υπό την ιδιότητά μου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών και όχι σαν πρόεδρος της Ζενεγάλ. να τονίσω τέσσερα στοιχεία. Μη αναφερόμενο στις τεχνικές λεπτομέρειες του πακέτου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ανάγκη διεθνούς συνέπειας και ισότιμων συνθήκων. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αξανόμενο κατακαιρματισμό του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου λόγω πολιτικών αλλαγών, κυρίως της ΕΠΑ αλλά και με την προπτική του Brexit που αυξάνει την τάση. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να συγκρατηθούμε από την επιδίωξη διεθνών συμφωνιών. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λόγω πραγματικότητας. Θα πρέπει να αποφύγουμε περιπτώσεις όπου η Ευρώπη δίνει ατελείς προτάσεις, όπως στην περίπτωση εξηγίας των τραπεζών. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε τα μαθήματά μας, κυρίως της αναθεώρησης του trading book, που δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα από την ομάδα της Βασιλείας. Πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστούν στις μεγάλες δικαιοδοσίες, όπως τις είπα. Υπάρχει σύγχυση. Άρα η αύξηση του κεφαλαίου, όπως εκτιμάται από τη Βασιλεία, διπλασιάστηκε από τον Εύριο του 2016 και το Φεβρουάριο του 2017. Το Νοέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόταση βάσει του πλαισίου της Βασιλείας. Και τώρα, το Φεβρουάριο του 2017, οι υπολογισμοί της Βασιλείας δείχνουν ότι φτάνουμε σε 80% αύξηση των κεφαλαίων. Είναι σημαντικό όταν πρέπει να σκεφτούμε στατηγικά την κατεύθυνση ακολουθήσουμε για την αγορά κεφαλαίων στην Ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειες του Brexit. Αυτό είναι το όλο υπόβαθρο. Οπότε ζητούμε από την Επιτροπή να αναβληθούν οι συζητήσει για τα OTP μέχρι το ότου υπάρχει ασφάλεια ε, και σαφήνεια σε επίπεδο ρυθμιστικό. Μετά η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να μεταφραστεί σε πραγματικότητα συνετή διαχείριση. Οι τράπεζε δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμα ένα πλήρω ολοκληρωμένο τραπεζικό σύστημα. Οι ευρωπαϊκέ τράπεζε αντιμετωπίζουν συμπληρωματικά κεφαλικέ απαιτήσει ε, και, και διαφορέ από νομοθεσία τα κριτήρια για εξαιρέσει όσον αφορά απαιτήσει, ρευστότητα κεφαλαϊκέ απαιτήσει έχουν επεκταθεί. Είναι ακόμα περιοριστική η όρη για είναι πρακτικά εφαρμόσιμο. 50% εγγύηση χρηματοδότηση για την ίδια χρηματοδότηση. Αυτό δεν αφαιρεί ότι το SSM και το ρυθμιστικό πλαίσιο έχουν ωφέλη. Η Ευρωζώνη είναι η δική μα εσωτερική αγορά και πριν να δούμε τι γίνεται μεταξύ συναλλαγών των διαφόρων πιστοτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να εφαρμοστούν και στου φορεί τη Τραπεζική Ένωση. Μετά πρέπει να δούμε ποια είναι η σημασία ε, ταχύων μεταρρυθμίσεων. Η ιεράρχηση των πιστωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά έχει θέσει την ιεράρχηση των πιστωτών σε ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο για να γίνει ταχεία εξέταση αυτού και να γίνει έγκαιρη η ε, υιοθέτηση αυτού. Γι' αυτό ο τομέα θα πρέπει να δει ποια είναι τα χρέη και να δημιουργήσει τα αναγκαία περιθώρια ταχαίω. Η Ομοσπονδία Τραπεζική υποστηρίζει την στέσπιση ενό σχήματο grandfathering για, ε, για τα στοιχεία παθητικού ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το IFRS 9 θα πρέπει το χρονοδιάγραμμα να καθοριστεί όσον αφορά τις διάφορες διατάξεις που προτείνονται θα πιστεύουμε επίσης ότι τα λογιστικά συστήματα που θα πρέπει να προσθούν τον Ιανουάριο του 2018 ζητούν επιταχυμένη συμφωνία του επόμενου μήνε, ώστε ε, τελικά να ακολουθηθούν οι κανόνε περί συνετής Τώρα σημασία της διαστάσεως αύξηση καινοτομία του πακέτου εμπεριέχει διάφορα ε, μέτρα για την αύξηση τη δανειοδοτική δυνατότητα των τραπεζών για να στηριχθεί ευρωπαϊκή οικονομία. Ελπίζουμε ότι εσεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εγκρίνετε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκταθεί η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια προτάσεω για να υποστηριχθούν επενδύσει για υποδομέ και να επιθυμίσω ότι στην Ευρώπη οι περισσότερε επενδύσει και τα διάφορα σχέδια μεταφορέ, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και νοσοκομεία χρηματοδοτούνται από τι τράπεζε. Θέλω να αναφερθώ επίση σε κάτι άλλο. Το πώ συμβάλλουν οι τραπέζε στην ψηφιοποίηση τη οικονομία τη Ευρωπαϊκή στην την ανάγκη οι να επενδύσουν σε ανάπτυξη λογισμικού για να παραμείνουν ε, ανταγωνιστικέ. Οι επενδύσει όμω είναι πιο δύσκολε ε, στην Ευρώπη από ό,τι στη ΣΥΠΑ για λογισμικό. Θεωρείται ότι είναι κάτι σαν εξοπλισμό στη ΣΥΠΑ το λογισμικό. Εν συμπεράσματι, θα ήθελα να αναπηχήσω το μήνυμα του Αντιπροέδρου Ντεμπόσκη ότι αναθέτησε το πακέτο για τη μείωση των προβλημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμμορφωθούν στι διαφόρες ιδιαιτερότητε του τραπεζικού τομέα της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της Ευρώπης, εν σειρά σα, να πετύχετε σωστή ισορροπία, να αποφύγετε επιβλαβείς αντίχτύπου στην πραγματική οικονομία και να αναπτύξουμε ένα βιώσιμο πλαίσιο για τις συμμετοχικές υπηρεσίες στην Ευρώπη που θα είναι κάτι επωφελίας για όλες τις οικονομίες μα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις διατάξεις αυτές, σειρά και αρτιτού Και να επιταχύνουμε. Επόμενος ομιλητής, Ανδρέας Τρέχλερ, που είναι ε, πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Erste Group Bank. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται όντω για το Group Este. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας το Este εδώ, στο κέντρο της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό για μας που είμαστε από αλλού, να συναντιόμαστε με ομολόγους μας από τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Έχω ένα μακρύ κατάλογο ε, από, τους, το προσωπικό του συναδέλφου μου για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να σας αναφέρω όσον αφορά τη ρύθμιση του ΤΙΛΑΚ, του MRL κλπ. Όμως, είμαστε από τη μεγαλύτερη τράπεζα σε έξι χώρες, θα τις ξέρετε. Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία, μεταξύ άλλων. Οι χώρες μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικές εποπτικές αρχές. Κάθε τόσο έχω την χαρά να συναντηθώ με κάποιον από τους πελάτες μου και με τους ανθρώπους που μας χρηματοδοτούν. Συνήθως όμως είμαι με ρυθμιστές και πολιτικούς. Πάντως χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Δεν θα σταθώ στις σημειώσεις μου γιατί θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ καλό. Φροντίστε να το ολοκληρώσετε. Δεν με ενδιαφέρει το πώς θα το ολοκληρώσετε, αλλά ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις αυτές και εγώ θα δεχτώ οτιδήποτε αποφασίσετε. Κάντε το όμως και μην το αλλάξετε τα επόμενα δέκα χρόνια, για να ξέρουμε ότι θα είναι σταθερό. Αυτό είναι το μόνο που έχω να σας ζητήσω. Όμως έχω να σας ζητήσω και κάτι ακόμα. Και σας παρακαλώ, προβληματιστείτε για το τι έχετε κάνει και για μας. Οι ρυθμιστές, οι πολιτικοί, οι τράπεζες στην Ευρώπη είναι πράγματα χρήσιμα. Και είτε εξυπηρετούν το σκοπό που θα έπρεπε όλοι να εξυπηρετούμε, δηλαδή ε, να δημιουργούν ευημερία για όλους στην Ευρώπη, μπορώ να σας πω από τη δικιά μου την εμπειρία ότι λειτουργούμε σε μια περιοχή της Ευρώπης όπου πολλοί κόσμος πληρώνουν 400-400 ευρώ το μήνα και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο αυτό να ε, βοηθήσει και εμείς στην περιοχή όπου βρίσκεται ο κόσμος αυτός να βοηθήσουμε να υπάρξει ευημερία. Και ο λόγος σε ένα βαθμό είσαστε εσείς οι πολιτικοί και σε ένα βαθμό είσαστε εσείς οι ρυθμιστές. Δεν μας διευκολύνεται τη ζωή για να δημιουργήσουμε ευημερία. Μιλάω για ε, το δανειστικό τμήμα. Αυτό είναι ένα. Μία από τις ε, συνέπειες ε, των όσων έχουμε ρυθμίσει είναι ότι καταστρέφουμε τις τράπεζες, γιατί τελικά οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν τίποτα πια σε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει ασφάλεια, ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει εγγύησεις και δεν έχει και κανέναν που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν εγγυητή. Έτσι δυστυχώς δεν έχουμε και εναλλακτικά μέσα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτά τα κεφάλαια κινδύνου δεν είναι τίποτα τελικά. Είναι ψίχουλα. Χρειαζόμαστε δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια και ξανά δισεκατομμύρια προκειμένου να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα άλλο πέρα από τη δουλειά τους, τη σκληρή δουλειά τους και την πίστη τους στο μέλλον και δεν υπάρχει καμία κατηγορία τελικά για δανεισμό πια. Αν αυτό δεν αλλάξει, τότε η Ευρώπη θα βρεθεί σε τεράστιο μειονέκτημα απέναντι σε άλλες περιοχές του κόσμου που αυτό γίνεται. Και γιατί? Γιατί η Ευρώπη είναι μια κοινωνία η οποία είναι προσανατολισμένη στο τέλος, στο θάνατο. Υπάρχουν ε, χώρες όπως είναι η Ελβετία που δεν είναι ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο που θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου να είναι, που τα έχουν καταφέρει. Οι άλλε όχι, ούτε η Γερμανία, ούτε η Σουηδία, ούτε η Ισπανία αρκετά. Αφήστε πια για τη δικιά μου χώρα και περιοχή. Δεν υπάρχει κεφαλαϊκή αγορά και δεν πρόκειται να υπάρξει κεφαλαϊκή αγορά τα επόμενα 50 χρόνια. Οπότε ποιο νομίζετε ότι τελικά θα χρηματοδοτήσει τι καινούργιε επιχειρήσει τις startups. Δεν υπάρχει κυβερνητική αγορά, δεν υπάρχουν οι επενδυτές. Οι τράπεζε αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερε δυσκολίε να δανείσουν. Οπότε τι θα γίνει. Αυτά από την πλευρά του δανεισμού. Τώρα, από την πλευρά τη δημιουργία πλούτου για τον κόσμο. Για τον κόσμο που βγάζει το πολύ χίλια ευρώ το μήνα. Πόσα θα βάλουν, 50 στην πάντα. Συλλογικά λοιπόν ως ρυθμιστές πολιτικοί και τράπεζες έχουμε αφαιρέσει από μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων την ικανότητα να έχουν χρήματα χωρίς κίνδυνο. Κοιτάξτε αυτό το πίνακα που σας ε, δείχνω και προσπαθήστε να το συγκρατήσετε. Δεν συνειδητοποιούμε πόσο τραγική είναι η αλλαγή η οποία έχει λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αφαιρέσει από όλους τους Γερμανούς, τη μεσαία τάξη, τους Αυστριακούς, ε, Τσέχους, ε, Ολλανδούς, τη μεσαία τάξη δηλαδή, το δικαίωμα να μπορούν να βάλουν στην πάντα κάτι από αυτά που κερδίζουν με τη δουλειά τους. Αν ε, επενδύσετε σε γερμανικό ομόλογο θα χάσετε, σε αυστριακό ε, αξιόγραφο θα χάσετε κλπ. κλπ. Δεν μπορείτε δηλαδή πια να επενδύσετε χωρίς υψηλό κίνδυνο. Δεν μπορείτε να βάλετε στην πάντα χρήματα γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από την απόδοση των χρημάτων σας. Τώρα λοιπόν, όπου μεγαλώνει μια γενιά που θα έχει μια εντελώς διαφορετική ιδέα για το τι είναι χρήμα, τι θα κάνουμε αν έχετε ασφάλεια, εγγυήσεις, μπορείτε να βγάλετε λεφτά από το τίποτα. Και αν έχετε χρήματα, πρέπει να είσαστε πολύ πλούσιος για να μπορέσετε να αναλάβετε τον κίνδυνο. Αλλιώς δεν μπορείτε να βγάλετε χρήμα. Αυτή είναι μια αλυσίδα λοιπόν. Είτε με τα TILAC e είτε με τα MRL δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, δεν αλλάξουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η είναι η επόμενη ομιλήτρια από την Τράπεζα Τρίοδος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, εκτιμούμε πολύ τη δουλειά που κάνετε για να γίνουν πιο ανθεκτικές οι τράπεζες και συμφωνώ ότι θα είναι χρήσιμο να ολοκληρωθεί αυτή η δέσμη μέτρων. Είμαστε εμείς διαφορετική τράπεζα, είμαστε ευρωπαϊκοί ε, και ασχολούμαστε και με τη διαχείριση επενδύσεων. 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε στοιχεία του ενεργητικού και 600 ε, πελάτες εξυπηρετούμε. Χρησιμοποιούμε τα χρήματα της αποταμίευσης για να επενδύσουμε σε βιώσιμες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ε, στεγαστικά δάνεια και ε, το δικό μας ποσοστό ε, είναι γύρω στο 20%, οπότε δεν ήταν κάτω από 13,8%. Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να δημιουργήσουμε μια οικονομία κοινωνική, ευφυή και βιώσιμη. Η, τρίοδος, η Τράπεζα Τρίοδος επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι απαραίτητο να υπάρχει η σχετική υποδομή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επικροτούμε επίσης ότι ασχολείστε με την αναλογικότητα. Για να υπάρχει βιώσιμη υποδομή ε, ε, θέλουμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας ε, διότι το να ελέγξουμε τον κίνδυνο σε τέτοιου είδους έκθεση ε, ευθυγραμμίζεται με την δική μας ε, πρόταση και πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική και περιβαλλοντική πτυχή. Με πιο αυστηρά κριτήρια για, τη του κινδύνου μπορούμε να ε, αιτιολογήσουμε την μείωση του κινδύνου. Εμείς από τη φύση μας βρισκόμαστε πολύ κοντά στους πελάτες μας και γι' αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητες στους παγκόσμιους ε, κλειδονισμούς. Ε, θέλουμε οι άνθρωποι να ασχολούνται και με την ε, μακροπρόθεσμη απόδοση των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν μειώνουμε το ποσοστό κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο μας και έχουμε και έναν παράγοντα υποστήριξης για τις μεγάλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φροντίζουμε λοιπόν να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τρόπο βιώσιμο, με κριτήρια αντίστοιχα με αυτά της υποδομής, αλλά που είναι προσαρμοσμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι η αναλογικότητα ποτέ δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο εισβάρος της προληπτικότητας και της δέουσας επιμέλειας και ξέρω ότι και ο κύριος Γκίκολτ ε, γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αναλογικότητα και θα είναι χρήσιμο για μας εάν αυτό αναφερθεί ρητά στον διάλογο με τον επόπτη, διότι πιστεύουμε ότι με το σωστό τραπεζικό τοπίο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τους συστημικούς κινδύνους. Είμαστε οργανωμένοι διαφορετικά και αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προκλήσεις από τις μεγάλες τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και ένας διάλογος μεταξύ των εποπτών που μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση για τις τράπεζες, διότι μερικές φορές στις έξι χώρες όπου έχουμε τηγατρικές βλέπουμε διαφορετική προσέγγιση. Μια άλλη πτυχή της αναλογικότητας ε, είναι ο ανταγωνισμός ε, ανάμεσα στα διάφορα είδη τραπεζών υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, λογοδοτούν με την προσέγγιση των ε, κανονικών τραπεζών. Για παράδειγμα, έχω εγώ ποσοστό κινδύνου 35% ε, για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ έχω πολύ χαμηλές απώλειες. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίζεται η σόφρον προσέγγιση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι μικρές ε, τράπεζες ε, μπορούν να είναι ανθεκτικές ε, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ειδική τραπεζική προσέγγιση τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη λογική σας πρόταση για τα στεγαστικά δάνεια που θα πρέπει να εξετάσουμε. Κρίσια Στίβ Μίλλερ, Finance Watch. Ευχαριστώ Πρόεδρε που καλέσατε την, ε, τον φορέα μου για να μιλήσει. ορίζουμε το πακέτο της τράπεζας, συμπεριλαμβάνει διεθνείς προδιαγραφές που είναι σημαντικές και τις συμπεριλαμβάνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στις υποθέσεις που βασίζουν τις προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, παρά κάποια πρόοδο πετεύθη, το κεφάλαιο των τραπεζών δεν έχει αποκατασταθεί σε ασφαλή επίπεδα. Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σωμές έχει περίπου 1-3 ευρώ ε, κόκκινων δανείων προς απορρόφηση. Για αυτού και άλλους λόγους οι ευρωπαϊκές Τράπεζε εξακολουθούν να είναι πιο χαμηλά κεφαλοποιημένε από τις περισσότερες ε, τράπεζε σε άλλες οικονομίες, σημαντικέ οικονομίες. Δεύτερον, οι κανονισμοί για το κεφάλαιο των ε, τραπεζών δεν επιβραδύνει την οικονομία η, η διάθεση πιστώσεων από τις τράπεζες δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, τόσο μεγάλο πρόβλημα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπου υπάρχουν λήψεις ε, πιστώσεων αυτό σε δομικές, ε, δομικά προβλήματα όπως τα μη αποδοτικά δάνεια. Αυτό που ισχύει είναι ότι καλά κεφαλοποιημένες τράπεζες χρηματοδοτούνται υπό καλύτερους όρους και είναι πιο πιθανό να μπορούν να δανοδιωτούν την πραγματική ονομία. Τρίτον, το πρόβλημα ότι οι τράπεζε είναι πολύ μεγάλε για να χρεοκοπήσουν δεν έχει ακόμα λυθεί. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία κρίση, οι πολίτε για μία ακόμη φορά αντιμετωπίζουν το λογαριασμό για δεκάδων δισεκατομμύριων για να στηρίξουν τράπεζε που κλονίζονται. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η εξυγίανση όπω πρέπει. Είναι οι συστημικέ τράπεζε να μπορούν να είναι σταθερέ και να παρέχουν φερεγκαιότητα. Θα πρέπει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα να γίνει υγιές και κερδοφόρο για μία ακόμη φορά, χωρίς να χάσουμε ανταγωνιστικότητα και επικοινομορφία. Οι τράπεζες πρέπει να εστιαστούν ξανά επί ανταγωνισμού βάσει των στοιχείων ενεργητικού τους. Άρα, καλύτερα προϊόντα, καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες αποφάσεις δεν ε, να μην βελτιστοποιούν το κεφάλαιο. Υπάρχουν σχετικές συστάσεις στο πακέτο όσον αφορά την πρόταση. Το Finance Watch γνωρίζει το βάρος συμμορφώσεως για τους μικρότερους φορείς του τραπεζικού τομέα. Στόχος δεν θα πρέπει να είναι κατά την άποψή μας να πετύχουμε ε, λιγότερο λεπτομερή στοιχεία ή να υπάρχει λιγότερη διαφάνεια. Θέλουμε λιγότερες και απλούστες διαδικασίες αναφοράς. Καλωσορίζουμε αυτό προτείνει η EBA, δηλαδή αρμονισμένο εργαλείο συμμορφώσεως θα θέλαμε να δούμε πιο φιλόδοξη όμως προσέγγιση που θα οδηγεί σε ένα σημείο επαφής για αριθμιστικές αναφορές που θα λειτουργεί επί της εφάπαξ αρχής. Ε, θα θέλαμε να δούμε και εντολή για την EBA να αναπτύξει ενοποιημένο σύστημα για λογιστικά, για αριθμιστικά θέματα και για υποβολή αναφορών για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πιστεύουμε ότι ο προτινόμενος ορισμός των μικρών θεσμών θα πρέπει να είναι πιο διαφοροποιημένος και να συνδυάνει ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα αντικατοπτρίζει το καθεστώς SII, δηλαδή συνδυασμό απολύτων και σχετικών κριτηρίων μεγέθους και κριτήρια που σχετίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο του, του, του φορέα και το μοντέλο ε, του κινδύνου. Χρειάζεται πιο ενήμερη συζήτηση για την αναθεώρηση του καθεστώτος του πυλώνα 2 και των κατευθυντηρίων γραμμών αυτού. Οι κατευθείαν γραμμέ του πυλώνα 2 θεσπίστηκαν στην επο... και εφαρμόστηκαν από την ECB και την EBA το 2016. Με μία μονοκονδυλιά ε, υπάρχουν κεφαλικέ απαιτήσει στα πλαίσια του SSM και μειώθηκαν κατά μέσο όρο οι απαιτήσει κατά 23%. Το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει περισσότερα πώς να επικρίνει το κεκτημένο και θα πρέπει να βασιστεί σε στοιχεία Χρειάζεται ενδελεχής αναθεώρηση τη ρυθμιστική πρακτική που τήθηκε πρόσφατα. Χρειάζεται και πλήρη αξιολόγηση συνεπιών πριν θετηθούν αυτέ οι πάρα πολύ σημαντικέ αλλαγέ που προτείνονται και πριν θεσπιστεί σχετική νομοθεσία. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα συνετή διαχείριση, η διαγραφή του άρθρου 103 του CRD, πρέπει να γίνει πριν αναθεώρηση των ε, μακροοικονομικών προσεγγίσεων για τη συνετή διαχείριση. Είναι κάτι που υποστηρίζουμε αυτό, αλλά πρέπει να ταιριάζει με ε, την κάλυψη κενών ρυθμιστικών. Καλούμε τους νομοθέτες να αναβάλουν τις προτινόμενες τροπολογίες του τμήματος 7 του κεφαλαίου 7 του CRD μέχρι ότου υπάρξει μια πλήρης πρόταση για εναρμόνιση μικρο- και μακροοικονομικών κανόνων για συνετή διαχείριση. Επίσης καλωσορίζουμε τη θέσπιση δεσμευτικού ε, ποσοστού μόχλευσης θα πρέπει όμως το 3% του ποσοστού μόχλευσης να δούμε ότι αντιστοιχεί στον ε, ελάχιστο ε, επίπεδο κινδύνου σύστημα, με το σύστημα Βασιλεία 3. Χρειάζεται υψηλότερο ποσοστό μόχλευσης για τις τράπεζες. Έχουμε και πλαίσιο TILAC, σημαντικό βήμα προόδου για την εξηγένση των τραπεζών, αλλά ακόμα και, πιο, και το πιο καλό πλαίσιο ε, είναι άχρηστο, δεν εφαρμοστεί όποτε χρειάζεται. Χρειάζεται αναθεώρηση λοιπόν του κανόνα για την προληπτική ανακεφαλοποίηση. Κάτι που εμποδίζει τη σωστή εφαρμογή του PRD. Δεν πρέπει να αποκλίνουμε από τα πρότυπα της Επιτροπής FSB και της Επιτροπής Βασιλείας, διότι θα υπονομευθεί η διεθνή συνεργασία για τις τράπεζες και θα υπονομευθεί και στις διαπραγματεύσεις η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το θέμα του ανταγωνισμού και της αντοχής των Ευρωπαϊκών Τραπεζών θα υπονομευτεί πιστεύουμε ότι ο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα δεν σε θέση που επιτρέπει σημαντικέ παραχωρήσει όσον αφορά τη μείωση των κεφαλουχικών απαιτήσεων που είναι δεσμευτικέ. Τελικά, καλούμε του νομοθέτε να αναθεωρήσουν τα διάφορα εμπόδια που υφίστανται όσον αφορά το καθεστώ εξυγίανση τη Βασιλεία, το καθεστώ BRD για την εξυγίανση των τραπεζών και θα πρέπει να εφαρμόζεται ασφαλώ και συνεπώ στο πλαίσιο αυτό για να διευκολύνεται η ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τους ευρωβουλευτές. Τρία λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Κάρας πρώτα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους μας τους ομιλητές που ήρθαν εδώ και που μας έχουν παρουσιάσει μια ευρία γκάμα απόψεων. Σε όλες τις ομιλίες που ακούσαμε σήμερα, τονίστηκε πόσο σημαντικό είναι η ρύθμιση για τις εκαθαρίσεις να συνεργάζεται στενά με την πολιτική. Αναμφισβήτητα, όπως έδειξε και η παρέμβαση του κυρίου Τράιχλ, Ε, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε επικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά την νομοθεσία μας. Έχουμε αντιπαραγωγική νομοθεσία. Η αναλογικότητα από μόνη της δεν αποτελεί λύση. Ούτε η παράταση της λύσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και γι' αυτό ρωτώ εγώ με τη σειρά μου. Στη ρύθμιση που είχαμε μέχρι τώρα, ποια ήταν τα δύναμα σημεία που μπορούμε να αλλάξουμε με την ε, νέα ρύθμιση. τι διορθωτικές κινήσεις μπορούμε να κάνουμε πέρα από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι αρκεί να αφαιθούμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη στις χώρες ε, της ε, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουμε ανάπτυξη της αγοράς. Η ρύθμιση αυτή θα αρκέσει και για τις χώρες αυτές και αν όχι, τι θα πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, όσον αφορά την αναλογικότητα, έχουμε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε ορισμό. Η υποβολή εκθέσεων από μόνη της μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους, αλλά επειδή έχουμε διπλή υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, το ότι υποβάλλει κάποιος μια έκθεση δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος απαλλάσσεται. Εσείς πώς βλέπετε την ιδέα ορισμού ή κριτηρίων για τα πιο απλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πώς βλέπετε το θέμα της υποβολής εκθέσεων και πώς μπορούμε να λύσουμε τις ασυμφωνίες στην ρύθμιση την νομοθετική και πώς βλέπετε την πρόταση για τυποποίηση ε, μιας πλατφόρμας δεδομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Πέντρο Σίλβα Περέιρα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας για τα όσα μας είπαν. Επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, περνάω αμέσως στις ερωτήσεις μου. Πρώτον, για την αναλογικότητα. Σήμερα το πρωί είχαμε τους ρυθμιστές. Κανείς δεν του ρώτησε μάλλον για τη διακριτική ευχέρεια, για το θέμα τη διακριτική ευχέρεια. Κανένα δεν του ρώτησε για το επίπεδο τη διακριτική ευχέρεια, ίσω γιατί φανταζόμασταν ποια θα ήταν η απάντησή του. Τώρα που έχουμε του διάφορου ενδιαφερόμενου, θέλω να ξέρω στο πακέτο αυτό το επίπεδο τη διακριτική ευχέρεια είναι υπερβολικό. Θα έπρεπε η προσέγγιση μας να είναι πιο πολύ βάση αυστηρών κανόνων, όπου το επίπεδο της ευελιξίας να είναι το αντίστοιχο. Πού θα έπρεπε να μειωθεί το επίπεδο διακριτικής ευχέρειας των αρχών ε, εξυγίανσης. Τώρα έρχομαι στην ε, αναλογικότητα. Έχει γίνει πρόοδος. Αναγνωρίστε το διοικητικό άχθος, συζητιέται το θέμα της συχνότητας, της ακρίβειας, granulation, συζητιέται το ποιες πρέπει να είναι οι απαιτήσει των αναφορών, αλλά όσον αφορά την ίδια την εξυγίαση, η στάθμευση των απαιτήσεων MRL πρέπει να οδηγήσει σε εξαιρέσεις, σε διαφοροποίηση για να λάβουμε υπόψη μας τις μικρές τράπεζες την φύση κάποιων ε, τραπεζών που να είναι αποταμιευτικές και που δεν εκδίδουν ε, χρέος. Θα ήθελα περισσότερα γι' αυτό από σας. Τέλος, όσον αφορά το θέμα αυτού του senior non-preferred debt, παλιό χρέος μη προτιμησιακό. Ένα από τα στοιχεία, από τα επιχειρήματα και τις ανησυχίες είναι ότι δημιουργώντας μια νέα τέτοια κατηγορία ε, δημοσίου χρέους, έχουμε την αίσθηση ότι μόνο αυτό το νέο χρέος θα ε, διασώζεται οι μέσες. Ρωτάω, είναι σωστή αυτή η εκτίμηση ή αντίθετα Πιστεύετε ότι αυτό το νέο είδος χρέους διευκολύνει αντίθετα και δεν περιορίζει την αποτελεσματικότητα του εργαλειου Μπέιλιν διάσωση της μέσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Άσλι Φόξ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας ε, για τις ε, παρουσιάσεις τους εδώ σήμερα. Ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Στάσερ όσον αφορά το διάστημα νομοθετικής ηρεμίας που ζήτησε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Εμείς οι πολιτικοί συνεχώς αλλάζουμε τους κανόνες και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να φτιάχνουμε νέους κανόνες και να τους αφήσουμε να κάνουν ε, ε, τη δουλειά που περιμένουμε από αυτούς. Κάποιες παρατηρήσεις ε, στο CRR αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ε, κάποια στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού μπορούν να θεωρηθούν ε, ότι αλληλοεξαρτώνται. Τα περισσότερα καλυμμένα ομόλογα όμως ε, δεν θεωρούνται ανεξάρτητα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και, κάτι, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασυμφωνία όσον αφορά το διάστημα λήξης Εάν έχουμε έκδοση δεκαετίας για ομόλογα υψηλής ποιότητας και αυτή η ασυμφωνία θα οδηγήσει σε ασυμμετρία λόγω της χρηματοδότησης που απαιτείται και της στάθμισής της. Όταν φτάσουμε λοιπόν σε διαστήματα χαμηλότερα του ενός έτους ή των έξι μηνών βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ασυμφωνία όσον αφορά το διάστημα λήξη ε, για τα ομόλογα αυτά. Εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντικό τα ομόλογα αυτά να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα διασυνδεδεμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για να μετριάσουμε αυτές τις ασυμφωνίες και τι άλλα μέτρα θα θεωρούσατε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφύγουμε τέτοια αποτέλεσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέγκας έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά αυτά που είπε και ο Ανδρέας, έχω να πω κάτι. Βέβαια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσεως Δημιουργήθηκε από κερδοσκοπική συμπεριφορά του χρηματοστικού συστήματος και αυτό οδήγησε στο να κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Αυτό οδήγησε σε μαζική χρέωση των ε, κρατών μελών, τεράστια χρέωση, και αυτό οδήγησε σε οδυνηρές συνέπειες για τη ζωή των πολιτών μας και των εργαζομένων μας. Άρα είναι κάπως ανησυχητικό να ακούω σε αυτή την αίθουσα ότι εμείς είμαστε οι ένοχοι ότι εμείς θέμε ότι τώρα πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα μέσω των οικονομιών μας, των αποταμιεύσεων μας. Είναι κάτι που άκουσα με κάποια δυσπιστία να αναφέρεται. Και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Το μη προτιμησιακό χρέος γιατί εκεί ε, υπάρχει ε, όφελος σε σχέση με τα άλλα είδη χρεών. Πώς θα δημιουργήσει, πώς θα λειτουργήσει αυτό στα διάφορα υποκαταστήματα των τραπεζών. Αυτό πώς θα επιληθεί ε, από πλευράς των πελατών. Δεν θα πρέπει να επικρατεί μυστήριο. Πρέπει να επικρατήσει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά το θέμα αυτό. Προς τον κύριο Ουντέα έχω ερώτηση. Όσον αφορά την ε, ολοκλήρωση των συμφωνιών Βασιλείας. Υποτίθεται ότι οι συμφωνίες της Βασιλείας θα έφεραν σε μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε σχέση με τις αμερικανικές. Στην πράξη αυτό πώς ισχύει, πώς επηρεάζεται η ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχει ο κίνδυνος τελικά να δεχθούμε μια εισβολή αμερικανικών τραπεζών. Και έχω και μία ερώτηση ε, για τον εκπρόσωπο της Finance Watch. Ακούσαμε κάτι για την προληπτική ε, ανακεφαλαιοποίηση. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας για τις αλλαγές του κανονισμού για μακροοικονομική συνετή διαχείριση, κυρίως τις αλλαγές όσον αφορά τον πυλώνα υπαριθμών 2 και για την εκπρόσωπο της ε, Τράπεζας Τρίοδος. Θέλω να την ευχαριστήσω πολύ για τα σχόλιά της, όμως όσον αφορά το θέμα του κινδύνου. Ε, ε, είναι μια τράπεζα που έχει μια θέση στην αγορά Σάμια τράπεζα που στηρίζει τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία υποδομών. Τι κάνετε για τη διαχείριση του κινδύνου, πώς λειτουργεί αυτό, πώς μπορείτε να χειριστείτε τον κίνδυνο για να σέβεστε τις προδιαγραφές που θέλουμε να εφαρμόσουμε μέσω αυτής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ, Σβέν Γκίγκολντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα έχω ερώτηση απευθυνόμαστε στην εκπρόσωπο της Τρίοδος Έχετε κάποιες προτάσεις στα πλαίσια του CRD και του CRR. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ότι το κλίμα και το περιβάλλον ή τα, οι κίνδυνοι ESG όπως αποκαλούνται αντικατοπτρίζονται καλύτερα. Αυτό που έθεσε η κυρία Περβάνς Περές στο, σαν ερώτημα στον προηγούμενο γύρο. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε κύριε Ράιχελ. Αυτό που περιγράψατε σαν αποτέλεσμα για την κοινωνική δανειοδότηση είναι κάτι ανησυχητικό. Ποιες προδιαγραφές θα θέλατε να αλλάξουν ακριβώς για να αποφευχθούν αυτές οι συνέπειες που περιγράφατε και δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να προβούσε ένα σχόλιο. Στην παρέμβασή σας υπήρξε μια μεγάλη αντίφαση. Είπατε καταρχάς μην αλλάξετε τίποτα σας παρακαλώ πια αμέσως μετά είπατε τι πρέπει να αλλάξουμε όλοι. Δεν υπήρξε συνέπεια. Πρέπει να το πω αυτό. Όμως ξεκολουθώ να πιστεύω ότι τίποτα από αυτά που κάναμε μέχρι τώρα ε, δεν διέπεται από τη διατήρηση της φύσης, την προστασία της φύσης. Δεν λέω ότι κάναμε τα πάντα. Καλωσορίζω η αδίποτε συγκεκριμένη πρόταση. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το καθεστώς σχετικά με αυτό. Πώς μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα χωρίς να υπονομεύουμε τη σταθερότητα. Τέλος, να πω και κάτι άλλο. Σε μια οικονομία της αγοράς δεν μπορούμε να έχουμε απόδοση ανευκινδύνου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πια. Και αυτό καθε αυτό δεν είναι ασφαλμένο, διότι σημαίνει ότι κερδίζεις κάτι χωρίς να δουλεύεις διαφορετικά και χωρίς να αναλαμβάνεις κάποιο κίνδυνο. Ξέρω ότι η εξαφάνιση του κέρδους, του περιθωρίου κέρδους, είναι κάτι δραματικό για το τομέα τον χρηματοστοτικών, αλλά είναι κανονικό σε μια οικονομία της αγοράς που είναι πλούσια σε κεφάλαιο. Τέλος, προς τον κύριο Σάτμαν Φάλης. Μπορείτε να μας να καταλάβουμε καλύτερα τον ορισμό της επιλεξιμότητας ε, για το μικρό αυτό τραπεζικό τομέα που είπατε. Είπατε ότι πρέπει να είναι μικροί θεσμοί και με μικρό κίνδυνο. Ο ορισμός σας όμως συμπεριέλαβε, από ό,τι κατάλαβα, και μικρότερους θεσμούς που αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους. Δεν κατάλαβα αν υπήρχε κάποια συνοχή στην πρότασή σας. Μπορείτε να μας δώσετε λεπτομερή κατάλογο αλλαγών που επιθυμείτε για να βοηθήσετε να επικρατήσει τελικά η αναλογικότητα στις προσπαθίες μας. Thank Σας ευχαριστούμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από άλλη πολιτική ομάδα να θέλει το λόγο. Για κάτι the έχουμε λίγο χρόνο. Εδώ, κύριο Σίγμαν. Και ο κύριος Χόκμαρ μετά. Δύο λεπτά, ο καθένας. Θα είμαι πολύ σύντομα. Θα ήθελα πολύ σύντομα να επανέλθω ε, στις προθεσμίες κοινοποίησης. Ε, δεν ακούσαμε πολύ, πολλές απαντήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να υποβάλλονται πάρα πολλά δεδομένα, παρόμοια, όχι όμως τα ίδια. Και το μεγάλο άχθος που προκύπτει από ε, τις εκθέσεις αυτές ε, που μοιάζουν μεταξύ τους ε, αλλά δεν είναι όμοιες, πώς μπορεί να μειωθεί. Δεν έχω την εντύπωση ότι οι τράπεζες έχουν συμβαστεί με τη λύση αυτή. Νομίζω ότι όλοι θα ήθελαν να απλοποιηθεί ο τρόπο υποβολή των δεδομένων και θα ήθελα οι επόπτε που βρίσκονται εδώ σήμερα να μου πούνε λίγα λόγια. Να μου πούνε αν θα μπορούσαν να φανταστούν για τέτοια λύση και αν όχι γιατί όχι. Ο κύριος Χόκμαρ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της εμπειρίας που έχουμε από την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγένση, την BRRD. Θα ήθελα δηλαδή σχόλια για το πώς βλέπετε εσείς τον καταμερισμό ευθυνών. Εποπτικές αρχές, αρχές εξυγένσης. Κάποιοι αποφασίζουν για το ΑΜΕΡΕΛ και άλλοι αποφασίζουν για το κατά πόσο οι απαιτήσει κατηγοριών είναι επαρκείς. Θα ήθελα λοιπόν μια πιο συνολική εικόνα. Ο καθένας το βλέπει από μια διαφορετική οπτική γωνία. Και αυτό μπορεί να δημιουργεί κάποια από τα προβλήματα που συζητήσαμε νωρίτερα που είπε ο κύριος Τρέχλ για μια συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης. Πού λοιπόν, πώς γίνεται ο καταμερισμός αυτός των ευθυνών, αυτό θέλω να ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ο κίνδυνος ότι τράπεζες που δεν έχουν αρκετό κεφάλαιο τιμωρούνται από κάποιες άλλες που έχουν υψηλό MRL. Ακριβώς γιατί ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα είναι από διαφορετική οπτική γωνία, οπότε δύσκολα συγκρίσιμα. Ωραία. Θα είναι μια μεγάλη αλλαγή, λέει ο Πρόεδρος, το να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Σωστή ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Χόκμαρ. Πρόεδρο, ωραία, δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο, στο ΚΑΤΣΔΙ. Συνεπώ. απαντήσεις από τους προσκεκλημένου μας, με την ίδια σειρά. Ο κύριος Σάκμαν ε, Φάλης πρώτα. Θα αρχίσω και μετά θα αφήσω το λόγο στον Φρέντερικ, μια που είναι εκείνο ο πρόεδρος της Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Εγώ θέλω να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση ναι, είναι πρόβλημα. Και υπάρχει το ζήτημα της μη καθαρής διάκρισης ανάμεσα στην εξυγίανση και τις εποπτικές δραστηριότητες. Βλέπουμε δηλαδή να, να υπάρχουν κάποια καθήκοντα που επικαλύπτονται μεταξύ τους. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων ε, μεταξύ των ε, μακρο και ε, οικονομικών αρχών εξηγένσεις. Εδώ είναι και οι συνάδελφοι, δεν θα τα πω εγώ. Πάντως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή εξέδωσε τις προτάσεις της βάσει κάποιων προτύπων. Θέλει ισχυρές απαιτήσει αναφοράς, αλλά θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να ασχολείται λίγο και με τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις δραστηριότητε και τη διαμεσολάβηση να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στην εφαρμοστική και νομοθετική εποπτεία. Κάτι το οποίο δεν έχουμε. Και σε ένα βαθμό το πακέτο οδηγία κανονισμός για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις έχει να κάνει με αυτό. Εγώ θα ήθελα να έχουμε σαφή διάκριση ευθυνών και να υπάρχει και απλοποίηση. Αυτό το χαρακτηριστικό να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Είναι πολύ πιο σημαντικό σήμερα από παλιότερα και δημιουργεί τεράστια απογοήτευση. Να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διάφορες λειτουργίες σε έξι χώρες και τελικά να έχεις δέκα επόπτες. Και επιπλέον έχουμε και άλλους τοπικούς ε, ελεγκτές εγώ ευχαρίστω να έχω έναν επόπτη και μία αρχή εξυγίανση και να συνομιλώ με μία αρχή. Άντε με δύο ή τρει το πολύ, αλλά όχι παραπάνω, παρακαλώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς γι' αυτό και φτιάχνουμε την Τραπεζική Ένωση, έτσι, για να τα... Ναι, αλλά δεν την κάνετε λέει ο κύριος Στρέικλ. Έχετε 8 χρόνια τώρα που το παλεύετε. Κάντε το έστω του χρόνου να γίνει. Πρόεδρος, ε, αν σκεφτούμε από πού ξεκινήσαμε, το να καταλήξουμε σε μια ενιαία αποπτική αρχή, νομίζω ότι είναι μεγάλο επίτευγμα. Ε, παρακαλώ τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στα, ερωτηματικά, στα ερωτήματα σχετικά ε, με την εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη των ε, κανόνων. Καταρχάς, οι μεγαλύτερες ε, επιχειρησιακές δυσκολίες βρίσκονται στην κοινοποίηση, διότι στις, στους μικρούς οργανισμούς αποτελούν το 50% των διοικητικών τους δραστηριοτήτων. 100 εργατοέτη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το άχθος για τις ε, μικρές και μεσές ε, τράπεζες της Ευρώπης. Γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, για την εποπτεία. Το 99% των πληροφοριών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια έχουν να κάνουν με το 8% των ε, πεδίων που πρέπει να ε, συμπληρωθούν. Το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μόνο αυτό το 8% των πληροφοριών για να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε πραγματικές ελαφρύνσεις, χρειαζόμαστε υποχρεώσεις κοινοποίησης, αλλά μόνο εφόσον υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, κάτι που δεν υπάρχουν ε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, δεν χρειαζόμαστε τους πολύπλοκους ε, κανόνες ε, για την αμοιβή των υπαλλήλων τους για τις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις. Επίσης, τα συμβούλια αυτών των τραπεζών δεν έχουν πολύπλοκες δομές ή υποεπιτροπών με τα ίδια μέλη κλπ. Επίσης χρειαζόμαστε εκ των υστέρων ε, έλεγχο, όχι όμως αυτόν τον πολύπλοκο εκ των προτέρων έλεγχο που έχουμε προβλέψει. Ε, αυτά λοιπόν θα είναι εφηρμοσμένη αναλογικότητα, όχι ε, μια ρέλια της επιχειρήσης που τους ή είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες. Αναφέρθηκα ήδη στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Οι μικρές ε, επιχειρήσεις με περιορισμένο κίνδυνο ε, ε, θα πρέπει να απελευθερωθούν από τους κανόνες της Βασιλείας που ούτως ή άλλως έχουν διαμορφωθεί με στόχο τις μεγάλες τράπεζες που εφαρμόζονται όμως σε όλες τις τράπεζες στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι εις βάρος της σταθερότητας ε, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αντιθέτως, θα διευκολύνει ε, τις πιστώσεις προς την πραγματική οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Στερβοντέα. Να σχολιάσω κάποια από τα θέματα που εφήγησαν όσον αφορά την αλογικότητα. Ένα σχόλιο. Εξαρτάται πιθανότητα τις τράπεζες τελούμε υποποπτία του SSM στα τράπεζε και περνάμε από ένα γύρο του BCBS 239 υποβολή αναφορών και περιέζεται στι οδηγίε ε, που εποπτεύονται άμεσα το TSSM. Είναι πολύ ε, παχθέ ε, έργο όσον αφορά την εφαρμογή τη αναλογικότητας. Όσον αφορά την επαγγελματικότητα, δεν περιορίζεται το κίνδυνο στο θέμα του μεγέθους. Βλέποντας την τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να πούμε ότι σημαντικός αριθμός προβλημάτων σχετίζονται με σχετικά μικρές τράπεζες με πολύ απλά επιχειρηματικά μοντέλα. Δεύτερον, η προτίμηση των χρεών, των παλιών χρεών. Στη Γαλλία έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για τη δημιουργία νέας κατηγορίας εργαλείων. Πήγε πολύ καλά με τις αγορές. πολιτική μας δεν απολούμε άμεσα στους δικούς μας πολιτές λιανικής, αλλά στους ενδιάμεσους φορείς που είναι σε καλύτερη κατάσταση να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να τιμολογήσουν. Πήγαν τα πράγματα ομαλά και μπορέσαμε να έχουμε τη νέα κατηγορία μέσων πέρα από το βασικό α, κεφάλαιο. Έχουμε και τα επίπεδα 1 και 3, όπως γνωρίζετε. Τα θέματα της βασιλείας και τα μοντέλα. Για τη βασιλεία. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη βασιλεία 4 και το ενδεχόμενο πρόσθετης αναθεωρήσεως των όσων ήδη εξετάσατε. Αυτά που είπαμε είναι ότι ανησυχούμε ότι οι ίδιοι κανόνες και καμιά φορά κανόνες λανθασμένοι εφαρμόζουν σε πολύ διαφορετικά συστήματα που χρηματοδοτούν την οικονομία και διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης θα διηγούσαν διαφορετικέ διαφορετικές συνέπειες. για τα στεγαστικά δάνεια, κάτι που αφορά όλους, είτε μικρές τράπεζες ή μεγάλες τράπεζες που ασχολούνται με στεγαστικά. Στη ΣΥΠΑ έχουμε δύο σκούπες που σαρώνουν Φένι Μέι και Φρέντι Μάρκ. Η Φάνι Μέι και Φρέντι Μάρκ που στηρίζονται από την κυβέρνηση και τροφοδοτούν στα στεγαστικά δάνεια. Και εμείς έχουμε στον ισολογισμό μας τα στεγαστικά δάνεια στην Ευρώπη είπε μακρόν. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για δύο διαφορετικά συστήματα, αλλά οι ίδιοι κανόνες δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο λόγω των διαφορών. Και γι' αυτό πρέπει να διαμορφωθούν σωστά οι κανόνες και έχει σημασία αυτό σε ένα περιβάλλον όπου οι τράπεζε είναι η βασική πάροχη χρηματοδοτήσεω της οικονομίας. Δεύτερον, συζητήσαμε εκτενώς και την εξειδικευμένη χρηματοδότηση. Ένα παράδειγμα γνωστό. Στην αρχή της πρόταση θέλαμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιο δάνειο μέσω εγγυήσεων ε, για τα αεροπλάνα. Μια αεροπορική εταιρεία. Οπότε εγγύηση είναι το αεροπλάνο. Πρέπει να, για αεροπορική εταιρεία να παραπλησιάσουμε επί εννέα ε, το ποσό ή τη χρηματοδότηση ε, για την αεροπορική εταιρεία. Και ένα δάνειο με εγγύηση που έχει εγγύηση αεροπλάνο θα πετούσε μεγαλύτερο κεφάλαιο από ένα δάνειο που δίνεται σε αεροπορική εταιρεία άμεσα χωρίς συγκεκριμένη εγγύηση εκτές από κάποια μοντέλα αεροσκαφών. Η αγορά των αεροσκαφών είναι σχετικά ρευστή. Έχει ρευστότητα. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε όλε τι συνέπειε. Και γι' αυτό λέμε στη Βασιλεία 4 ότι η Βασιλεία 4 θα έχει σημαντικότατε συνέπειε εάν δεν υπάρχει σωστή προσέγγιση και οικοδόμηση. Και γι' αυτό είναι καλύτερο να μην έχουμε συμφωνία καμία παρά κακή συμφωνία. Αν έχουμε μια καλή συμφωνία, γιατί όχι όμω. Για τα μοντέλα. Τι είναι τα μοντέλα προσπαθούμε, είναι ένας τρόπος να δούμε αποτελεσματικά τι είδου κίνδυνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, τι ίδιο πίστοση μπορεί να έχουμε, λαμβάνοντα υπόψη παρελθούσε εμπειρίε, τι απώλειε έχουμε ζήσει μέσω του κύκλου σε καλέ και κακέ εποχέ και να λάβουμε υπόψη αυτά σε ένα μοντέλο για τον υπολογισμό κεφαλαίου για το μέλλον. Υποστηρίζουμε αυτή την εκ των προτέρων μεθοδολογία, είναι πολύ σημαντική για μα γιατί έτσι εξετάζουμε εμεί τον κίνδυνό μα να πω ότι το SSM θα προσπαθήσει να αρμονίσει περαιτέρω αυτά τα μοντέλα για να εξασφαλίσουμε ε, ασφαλή προσέγγιση και να παίζουμε τα μοντέλα, αλλά σεβόμεθα τη σωστή μεθοδολογία. Τέταρτον, δεν έχω απάντηση στην ερώτηση που ετέθη για το SSF. Σε αυτό το κείμενο ξεπερνάμε αυτό το θέμα. Πρέπει να εξεταστούν διάφορα τράπεζα για το ποσοστό μόχλευσης. Πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως για να είναι λογικά. Για κίνδυνο, για ρευστότητα. Και μέσω της ερωτήσεως είδατε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Είναι περίπλοκοι οι κανόνες για το LCR, το ποσοστό ρευστότητα, το ποσοστό κεφαλαίου, το ποσοστό μόχλευση και όλα αυτά είναι πάρα πολύ περίπλοκα για να βρούμε σωστή ισορροπία μεταξύ όλων αυτών. Χρειάζεται όμω μια συνέπεια με την αντιμετώπιση του κινδύνου και με την ε, όλη διαχείριση του θέματος. Ευχαριστώ. Σαμπίν Τίμερς Γιάνσεν. Ωραία. Δύο ερωτήσεις θέλω να απαντήσω για τον δανεισμό και τον δανεισμό και δεύτερον πώς μπορούμε να καθορίσουμε την αναλογικότητα. Για το πρώτο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που πάντα κάνουμε κάθε φορά που πρόκειται για δανεισμό, κοιτούμε ποια είναι τα δανειστικά μας κριτήρια και διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετά περίπλοκα. Έτσι καλλιώς είναι τριπλά. Πρώτα πρέπει να δούμε κατά πόσο επιχειρηματία αντιλαμβάνεται καλά τη δουλειά του, αν πιστεύει στις ιδέες του και αν θα μπορέσει να τις κάνει να λειτουργήσουν. Άρα έχει να κάνει με την ίδια την προσωπικότητά του. Δεύτερον, εξετάζουμε πώς στηρίζεται από την τοπική κοινότητα, αν ο περίγυρός του στηρίζει την ιδέα του. Είτε πρόκειται για κοινωνικές, περιβαλλοντικές εξελίξεις, αλλαγές, αν όλα αυτά ε, είναι εφαρμόσιμα στο χώρο που βρίσκεται και τρίτον κατά πόσο θα είναι σε θέση να το κάνει να λειτουργήσει, αν αντιλαμβάνεται τι λεπτομέρειε και αν θα μπορέσει να έχει ένα λογικό κέρδο από τη δραστηριότητα αυτή. Εμεί πιστεύουμε ότι εξαρτώντα από αυτά τα τρία δανειστικά κριτήρια διασφαλίζουμε ότι τελικά έχει πάντα να κάνει με κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον για την κοινωνία. Και μόνο όταν τα κριτήρια αυτά καλύπτονται αρχίζουμε την αξιολόγηση κινδύνου ποιοτικά, ποσοτικά μέτρα και βέβαια όσο καλύτερα κάνουμε την αξιολόγηση κινδύνου, τόσο χαμηλότερη είναι και η κεφαλιακή απέτηση. Οπότε είναι ένας, πιστεύω, κατανατός εύκολος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, όταν μιλάμε για την αναλογικότητα. Πάντα είναι ένα περίπλοκο θέμα και έχει να κάνει με πολύπλοκους χώρου. Συνήθως μιλάμε για τις πιο μικρές ε, τράπεζες έχουμε λιγότερο προσωπικό στα γραφεία για να κάνουν τη δουλειά. Και για μένα αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει θα ήταν αν είχαμε πραγματικό διάλογο με τις αρμόδιες αρχές για το πού εφαρμόσουν την αναλλαγικότητα. Αυτό να φαίνεται πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή να μην πάει κάποιο να σε τσακώσει ότι ξεφέγγισε από τους κανόνες, αλλά να είναι αποφελής η δουλειά σου. Ίσως τα έπρεπε και εμείς να το δούμε, να είναι κάτι το οποίο θα μπει στην οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Οι ε, διάφοροι έλεγχοι, εξωτερικοί κτλ. είναι ενδιαφέροντες, αλλά δεν θα έπρεπε να προβλέπονται και τελικά να μην γίνονται. Και δεν θέλω να μιλάμε μόνο για κεφαλικά επίπεδα, γιατί η αναλογικότητα δεν θα λειτουργήσει τότε. Η συγκέντρωση δεδομένων θα έπρεπε να παίζει λιγότερο. Νομίζω ότι μας βοηθάει πολύ να έχουμε τις αναφορές, γιατί αυτό βοηθάει να καταλάβουμε την επιχείρηση του άλλου. Αλλά βλέπετε, έχουμε δύο που δουλεύουν στο γραφείο για αυτό το θέμα και είναι πολύ δικευμένοι, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά ε, τα καθήκοντά τους, αλλά τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξετάσουν χιλιάδες σελίδες ρύθμισης. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο πώς θα λάβουμε υπόψη μας την αναλογικότητα. Σε αυτό θα μπορούσατε ίσως να βοηθήσετε. Ευχαριστούμε. Χριστιαν Στιφ Ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις που απευθύνατε σε μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την προληπτική ανακεφαλοποίηση. Ποια είναι η άποψή μας πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι κατ' ουσίαν δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, ρητά μια ρήτρα διαφυγής. Πιστεύουμε ότι η αρχή αυτή αντίκειται ε, στον βασικό στόχο του BRRD. Έχουμε το πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι οι απώλειες απορροφούνται από τους πιστωτές που είναι καλύτερα σε θέση να τις χειριστούν, δηλαδή επαγγελματικοί οργανισμοί στο βαθμό που ε, τα μέσα κινδύνου καταλήγουν ε, σε λιανικούς επενδυτές που δεν μπορούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα της λάθος πώλησης και στο μέλλον θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε αυτούς τους μικρούς επενδυτές. Για παράδειγμα, τα ομόλογα 81 ε, μάλλον δεν ενδείκνυνται για τέτοιους επενδυτές. Επίσης, όσον αφορά την μικροπροληπτική και την μακροπροληπτική εποπτεία, τα μακροπροληπτικά πρότυπα θα πρέπει να τα καλύψουμε με αρμονισμένο τρόπο. Μας ανησυχεί όμως διότι από τη μία οι εποπτικές αρχές ήδη έχουν ασχοληθεί με τις μικροπροληπτικές υποχρεώσεις και τώρα ο νομοθέτης προτείνει σημαντικούς περιορισμούς στην ελευθερία των ρυθμιστών να ασχοληθούν με ιδιαίτερες κατηγορίες κινδύνου. Ταυτόχρονα, σε μακροπροληπτικό επίπεδο, και σας παραπέμπω σε πρόσφατη ε, μελέτη του ESRD. Ε, το τοπίο είναι πολύ ε, ανομοιόμορφο και αναθεώρηση του μακροπροληπτικού πλαισίου βρίσκεται καθοδόν. Εμείς πιστεύουμε ότι και οι δύο πλευρές και το μικροπροληπτικό και το μακροπροληπτικό πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο και εναρμονισμένο τρόπο. Όσον αφορά την αναλογικότητα, συμφωνούμε με πολλά από όσα υπόθηκαν όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για ελάφρυνση του άχθους. Αλλά είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε πρόταση για την απλοποίηση του άχθους θα οδηγήσει σε ελάφρυνση της μακροπροληπτικής εποπτείας. Το MRL e εξαρτάται από το σχέδιο εξυγίανσης που προβλέπουν οι αρχές για κάθε μεμονωμένη τράπεζα. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρξει εξυγίανση αλλά γίνει η δεν χρειάζεται ε, να εφαρμόζονται τα MRL, e οι ελάχιστε απαιτήσει ε, ίδιων κεφαλαίων. Σα ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ bail-in και του burden sharing διότι λέγατε ότι ο καταμεσμός του βάρους το, το, το, το κάλυπτε αυτό. Πρέπει να υπάρχει αυτή η διαποροποίηση όμως μεταξύ bail-in και του burden sharing. Δεν συμφωνώ με σας αυτό. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν τους εποπτικούς φορείς. Αν μας δίνει διερμηνείς λίγο χρόνο ακόμα, ένα σχόλιο για το MRL μπορώ να κάνω πριν απαντήσουν οι εποπτικοί φορεί, διότι είχαν χρόνο να μιλήσω. Αλλά δίνετε το δρόμο στον εαυτό σα άμεσα, αλλά ένα λεπτό, έτσι, διότι ήδη απαντήσατε. Για το MREL, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε, είναι καλό σημάδι διάκρισης μεταξύ εποπτείας, εποπτικών δραστηριοτήτων και ε, εξυγίανσης. Για το άλλο που αναφέρθηκε δεν υπάρχει σαφήνεια, πρέπει να επικρατήσει σαφήνεια. Υπάρχει τεράστιο αντίκτυπο στο επιχειρηματικό μοντέλο αν έχουμε πολλαπλά σημεία εισόδου ή ενίο σημείο εισόδου και δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις σε αυτού. Εάν δεν έχουμε πολλαπλά μια εισόδου σαν φορείς έχοντας έξι ισχυρέ τράπεζες λιανικής δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι και αυτό έχει σημαντικές συνέπειες όσον αφορά το μοντέλο. Και όσον αφορά αυτό το θέμα, η εξυγίανση και η εποπτεία θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη άποψη και να προβαίνουν σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση και άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να απαντήσει. Ανδρέα Ανρία, κοιτάξτε αν επιτρέπετε το ερώτημα του Πίτερ Σιμών για το θέμα της αναφοράς να τονίσω για τη συχνότητα, συμφωνώ με την Τανιέλ το θέμα της συχνότητας κυρίως όσον αφορά την έκθεση ρευστότητα, οι εποπτικοί φορείς δεν μπορούν να περιμένουν ένα χρόνο μέχρι να ξέρουν ποια είναι η θέση ρευστότητα της τράπεζας αν νομοθετική απέτηση είναι συχνότητα ενό έτους το αποτέλεσμα θα είναι πιο εντατική επιτόπια εξέταση μεγαλύτερο βάρος αλλού υπάρχουν τομείς όπου δεν μειώνουν τις απαιτήσει Ήδη πετύχαμε μεγάλη συνέπεια στον αφορά το κοινό πλαίσιο αναφορών. Πρέπει να ξέρουμε τι παράγει ακόμα το θέμα του βάρους αναφορών. Δηλαδή, πέρα στο κοινό πλαίσιο αναφορών, με το SSM και το SRB, έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα. Οι φορεί ενημερώνουν το SSM και το SSM ενημερώνει εμά ή το SRM. Υπάρχει ολοκλήρωση. Αυτό που δεν λειτουργεί είναι ότι πέραν αυτού, πέρα από τις απαιτήσει αυτής κοινή ε, ενημέρωση, υπάρχουν άλλες απαιτήσει από τι αρμόδιες αρχές, ε, ε, συνετή, διαχείριση κλπ. Και δημιουργούνται απαιτήσει αισθητικά στοιχεία. Στη ΣΥΠΑ, αρχές δεκαετίας 80, έχουμε Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Εξέταση Χρηματοπιστικών Ιδρυμάτων, όπου υποχρεώνει στις αρχές να μαζεύονται και να συμφωνούν επί ενιαίων απαιτήσεων για υποβολή αναφορών και αυτές είναι οι μόνες απαιτήσει που επιβάλλονται σε μία αρχή που τις μοιράζει στους άλλους. Αυτή είναι η λύση. Αν μπορούμε να το θεσπίσουμε αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντική η πρόοδος. Για τις ευθύνε και λοιπά και τις απαιτήσει δεν ήταν μια εξαίρεση που προβλεπόταν στην έκθεσή μας, στις συστάσεις μας. Αν έχετε διαφορετικά χαρακτηριστικά χρηματοδοτήσεως και ενεργητικού, πρέπει να καλύπτετε το ποσοστό χρηματοδοτήσεως. Υπάρχει μια πρόταση για εξαίρεση. Σύστασή μας είναι να ταιριάζεται με το ρήφθο δοθεί στο MBA για τα κριτήρια που θα αφορούν αυτό το θέμα, τι ακριβώς εννοούμε πότε το παθητικό και το ενεργητικό αλληλεξαρτώνται και πώς εξισορροπούνται και όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο αυτό. Δανία Νου είναι οι δύο σημεία όσον αφορά εναρμονισμένη κατηγορία μη προτιμησιακού παλαιού χρέους υποστηρίζουμε και γενική προτίμηση καταθετών και αν θέλαμε να, να βοηθήσουμε τον Μπέιλιν ή να το κάνουμε πιο περίπλοκο τον Μπέιλιν, όχι, θέλουμε να βοηθήσουμε τον Μπέιλιν. Πιστεύουμε ότι η αρχή εξυγίανσης θα μπορεί ε, να, να χρησιμοποιήσει στον Μπέιλιν και τα άλλα εργαλεία που υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι σημαντικό για τους φορείς της λιανικής, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αξιώσεων αποζημίσεως και την αρχή σύμφωνα την οποία κανένας μισθωτής δεν πρέπει να βρεθεί σε πιο δυσχερή θέση. Άρα πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη εξυγίανση. Τώρα, ε, τα καλυπτόμενα ομόλογα και αντιμετώπιση στο FNSR συμφωνούμε με τη σύσταση της ΕΜΠΑ του Δεκεμβρίου του 2015 σχετική έκθεση σύμφωνα με την οποία μόνο εκείνα τα ομόλογα που περνούν μέσα από τους διάφορους φορείς θα πρέπει να προβλέπονται σε εξαιρέσεις NSFR. Όλα τα άλλα ομόλογα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα NSFR. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος. Επιτρέψτε μου να επανέλθω λίγο στο ερώτημα του κύριου Χόκμαρ για την επίδραση της εποπτείας και της εξυγίανσης από τη δικιά μας την πλευρά. Η υπόθεση είναι αυτή η ιδέα ότι εφαρμόζουμε μετά από το Σαββατοκύριακο της εξυγένσης. Πρόκειται για μια τράπεζα υποεκαθάριση. Και ναι, έχετε δίκιο ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο επίπεδο της αποδοχής που έρχεται από πλευράς της εποπτείας πριν το Σαββατοκύριακο και μετά το Σαββατοκύριακο. Γιατί τι θέλουμε εμείς να διατηρήσουμε τις βασικές λειτουργίες της τράπεζας και θέλουμε να της επιτρέψουμε να συνεχίσει τις δραστηριότητές της. Οπότε είναι κάποια υπόθεση που παίρνουμε εξάντε, και αυτό είναι το λεπτό, για το ποιο θα πρέπει να είναι το σωστό επίπεδο. Και αυτό με το TILAC υπάρχει η αναφορά του 16% που είναι δύο φορές 8% στην πραγματικότητα που είναι το ελάχιστο στο ΤΙΛΑΚ. Αρχίζουμε λοιπόν από τις προσδοκίες ε, της εποπτικής αρχής και φτιάχνουμε το MRAIL και είναι το ίδιο σε διεθνές ε, επίπεδο και στο μελλοντικό πακέτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το MPSP. Εδώ δεν μπορώ να επαναλάβω αυτό που υπόθηκε ότι δεν είναι από τις αρχές που αποφασίζει τη δραστηριότητα τραπεζική, αν πούμε ότι είναι MP από τη μία, SP από την άλλη, αυτό συμβαίνει γιατί είναι περίπλοκες οι δραστηριότητες και δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα από πλευράς εξυγίανσης. Όχι από πλευράς ισολογισμού, από πλευράς εξυγίανσης υπάρχει το πρόβλημα και αυτό είναι που προσπαθούμε να λύσουμε. Εσείς. Ναι, και εγώ για το MRL και τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις και πώς αυτά τα δύο λειτουργούν ε, μαζί, το πρώτο ο κύριος Χόκμαρ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ως προσωπικό κίνητρο, εγώ ως επόπτης θα ήθελα να έχω μια ισχυρή τράπεζα, δεν θέλω να διακινδυνεύσει η φήμη μου, ενώ οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να έχουν και αυτές το ίδιο κίνητρο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Να έχουμε τα ίδια επίπεδα MRL πριν και μετά το Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και γι' αυτό και αξίζει τον κόπο η συζήτηση, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω απάντηση. Τώρα για τα ενυπόθηκα ομόλογα, Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και ο βασικός λόγος που δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία στην Επιτροπή της Βασιλείας ακόμα είναι η βασική διαφορά στο κίνδυνο αμερικανικών τραπεζών με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό είναι που κάνει την τεράστια διαφορά και δυσκολία. Όμως για το τραπεζικό σύστημα θέλουμε να υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία κάποιου είδους αλλά αυτή είναι μια από τι μεγαλύτερε δυσκολίε για να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε η Λίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τα MRL, πρέπει να, έχουμε, να προσέξουμε περισσότερο το θέμα, να γίνει αξιολόγηση αντίκτυπου όσον αφορά τα κοινά του MRL κατά την περίοδο κατά την οποία θεωρητικά θα ζητούμε παρα, να επιβάλλονται παραπάνω προϋποθέσεις και προσπαθούμε να εκτιμήσουμε το σχετικό κόστος. Μέσω κοινή προσεγγίσεως των τραπεζών. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και ο μέσος όρος δεν σημαίνει τίποτα εδώ. Δεύτερο, η ιεράρχηση πιστωτών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί και να επιταχυνθεί η διευκρίνηση. Τρίτον, αναφέρθηκε το ότι επειδή έχουμε νέα αγορά και επειδή έχουμε τραπεζική ένωση σε χρηματοσωτικούς ομίλους θα υπάρχει το όφελος από τη συγκέντρωση δυνατός απορρόφησης απολειών και με τη ρευστότητα σε κάποιες οικονομίες. Αυτός είναι ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε. Για την ώρα, κακές εποχές, πρέπει να έχουμε το ίδιο επίπεδο ευθυνών δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικέ καταστάσεις για, τα και υποκαταστήματα να έχουν εστέρηση ρευστότητες και υπάρχει αντίκτυπος και δεν καλείται το αντίκτυπο σωστά μέσω καταλήλων εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να συστούμε σε εθνικά μέσα. Αν το κάνουμε αυτό, δεν θα είμαστε σε σωστό πλαίσιο για τη διαχείριση οικονομίας. Τέλος, IFRS 9 πρέπει να επιταχυνθεί η μεταβατική περίοδος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πότε και υπό ποιους όρους θα εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ και τώρα οι συγγητές μας. Κύριε Όκμαρκ. Uh, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις τους και για τις απαντήσεις που δόθηκαν σε διάφορα ερωτήματα. Νομίζω ότι ακούσαμε διάφορα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε στη συνέχεια. Για παράδειγμα, το πώς μπορούμε να καθορίσουμε το σωστό επίπεδο του MRL ε, συμπεριλαμβανομένου του ΤΙΛΑΚ καθώς ε, και το επίπεδο ιδίων κεφαλαίων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος ε, θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα αυτό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και εγώ να ευχαριστήσω θερμά όλους σας ε, για αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Με ενδιαφέρον ακούσαμε ότι η αναλογικότητα είναι ένα από τα θέματα κλειδιά με τα οποία ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτό που είπε ο κύριος Ενρία. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Θα πρέπει να προσέξουμε να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τι ήδη έχει συμβεί. Με χαρά θα παραμείνω σε επαφή με όλους σας ε, στη συνέχεια κατά την εκπόνηση των εκθέσεων ε, για το CRR και το CRD, τον κανονισμό και την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό το σεμινάριο αυτό. Τώρα λοιπόν έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσής μας ε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλή νομοθεσία.